Okay, well, I'm going to start anyway. Λοιπόν, θα αρχίσω έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε μερικούς ε, που θα φτάσουν αργότερα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αφού είμαστε και στη διαδικασία Meetings, then, uh... συνεδριάσεων των σκιωδών εισηγητών, ε, θα τα πούμε. Ε, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί είναι το υπαριθμό 9. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα και σε χρηματοπιστωτικές συμβάσεις. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις τροπολογίες και όπως γνωρίζετε όλοι σας, εγώ είμαι η συγγήτρια, έχω την τιμή αυτή. Μου το ανέθεσαν οι συντονιστές εν τη σοφία του στην απεριόριστη. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τα μέλη και τους σκιώδεις για τις τροπολογίες τους. Γενικά τις θεωρώ χρήσιμες για να πάμε σε μια καλή κατεύθυνση. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε συμβαστικές τροπολογίες που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε μια λογική θέση για την ψηφοφορία. Όπως σας έχω πει, χωρίζω σε δύο τμήματα την έκθεσή μου και ο δεύτερος γύρος των τροπολογιών καλύπτει κάποιους τομείς που δεν είχα συμπεριλάβει και καλύπτει και κάποιες συζητήσεις που έγιναν και με τους σκιώδες συγητές και εδώ στην Επιτροπή μας. Έχουμε ήδη συνεδριάσει και εγώ έχω κάνει ήδη κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις για να συγκεντρώσουμε πολλές τροπολογίες των συναδέλφων και να βοηθήσουμε να διευκρινιστεί η υπόθεση όσο και να απλουστευτεί. Τα νέα τώρα από το Συμβούλιο ποια είναι, θα αρχίσουν να εργάζονται επ' αυτού, αλλά μάλλον περί τα μέσα Φεβρουαρίου, όχι νωρίτερα. Είναι πολύ δύσκολο, μην πω, αδύνατο να φτάσουμε σε τριμερή διάλογο, αλλά τουλάχιστον να διαμορφώσουμε εμεί μια θέση και να τους τη δώσουμε να την κοιτάνε όσο θα δουλεύουν και εκείνοι όταν αρχίσουν. Προς το παρόν, θα πρότεινα περί τις 17-20 Φεβρουαρίου να ψηφίσουμε εμείς. Το έχουμε ήδη συζητήσει με τους σκιώδες και θα γίνουν και άλλες συνεδριάσεις την άλλη εβδομάδα. Προσπάθησα να κάνω νέες τροπολογίες και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα πούν και οι συνάδελφοι τα δικά τους και θα κάνω μια πρόταση. Έχω τροποποιήσει λίγο στο άρθρο 5.1 της ιδέας μου, στην τροπολογία 282 συγκεκριμένα, για να ε, συμπληρωθεί και από την ε, πραγματογνωμοσύνη της ε, ΕΣΑ ως προς το πεδίο εφαρμογής, η ΕΑΚΑ δηλαδή, ε, για τους δείκτες ε, ε, αναφοράς και για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Η ΕΣΜΑ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών, θα πρέπει να επιληφθεί. Συνήθως ο κόσμος Αυτά τα θεωρεί στο άρθρο 2 ότι πρέπει να υπάρχουν, αλλά εγώ θέλω και ε, ένα κατάλογο ή ε, μία έκθεση για τη διακυβέρνηση. Πάντα μας λένε ότι ναι, ναι, τα έχουμε αυτά τα ισοδύναμα και τους δείκτες, ιδιαίτερα για ομόλογα τρίτων κρατών, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος έλεγχος, ε, και όχι απλώς λεκτικός. Επίσης θέλω να ζητήσω από την ΕΣΜΑ, ΕΑΚΑ, να μας πει ποιες ε, ρυθμισμένες αγορές καλύπτονται από το REMIT. Δεν θέλω γενικές εξαιρέσεις έτσι ε, αδιάκριτες, πάντα να πρέπει να γίνεται μια διαβούλευση γιατί προσπαθώ κατά κάποιο τρόπο να ικανοποιήσω όλους εκείνους που θέλουν ευρία κάλυψη, αλλά να υπάρχει και κάποια στοιχειώδης εποπτεία χωρίς μεγάλους περιορισμούς, αλλά όχι τελείως ε, ανεξέλεγκτη όταν λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση προοδευτικής εισόδου στον κανονισμό ε, phased in. Το έχουμε ήδη ε, κάνει αυτό για κάποιες υπηρεσίες που αναφέρουν στοιχεία για τις τιμές, οίκους αξιολόγησης κτλ. Οι διαχειριστές λοιπόν θα πρέπει με ε, ε, πράξεις κάτω εξουσιοδότηση και άλλες να καλύπτονται. Στις συζητήσεις που είχαμε λοιπόν με τους σκιώδεις ηγητές, διεφανεί ότι ορισμένοι θεώρησαν ότι καλό θα ήταν στο άρθρο 2 να μπουν αυτές οι προσαρμογές που προτείνω για το πεδίο εφαρμογής και όχι στο άρθρο 5. Αυτό θα προσπαθήσω να το κάνω στις συμβαστικές τροπολογίες γιατί νομίζω ότι είναι σωστό. Για τους διάφορους ορισμούς τώρα, η μεγαλύτερη τροπολογία που έκανα ε, είναι ε, να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στα ρυθμισμένα δεδομένα και στα ε, δεδομένα αναφοράς. και ενδεχομένως ε, και δεδομένα ότι ε, στον ε, κανονισμό αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω αυτό στέλνει κάποια λάθος μηνύματα γιατί θέλουμε να εθαρρύνουμε την αγορά. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη ρυθμισμένη αγορά με στοιχεία και δεδομένα πιο ακριβή και πιο αξιόπιστα. Θα δούμε πώς μπορούμε να το προσθέσουμε αυτό όταν δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια. Ε, έχω αλλάξει και το όριο. Τα 500 δις ε, για το κρίσιμο ε, επίπεδο το έχω διατηρήσει, αλλά είναι δύσκολο να υπολογιστεί αυτό ως ποσό και μπορούν να υπάρξουν κάποιες ανομαλίες ή στρεβλώσεις η ΕΑΚΑ θα πρέπει εκείνη να ορίζει ποιο είναι το κρίσιμο όριο με βάση τις διεθνείς αγορές και να προτείνει ένα υποκατάστατο. Αλλά 500 δισεκατομμύρια είναι ένας αριθμός που δείχνει ένα, στέλνει καλύτερα ένα σαφές μήνυμα. Δεν χρειάζεται να τα μετράμε μέχρι τελευταίο ευρώ για ε, τα 100 δις και αυτό το κατόφλι για το βασικό ε, benchmark, ε, κριτήριο αξιολόγησης και αυτό το έχω κάπως αλλάξει για να έχουμε την ευκαιρία να οπλουστεύσουμε λίγο τα πράγματα. Θα ακούσω και τις δικές σας απόψεις για αυτό το θέμα. Θα ε, παρακαλούσα ε, να δεχθούμε οι διαχειριστές να διαπιστώσουν να δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους ή τα στοιχεία. Εξαρτάται τι οργανισμός είσαι. Αν είσαι ένας ε, οργανισμός αναφοράς τιμών δεν έχεις πρόβλημα να ε, δημοσιοποιείς και τη μεθοδολογία σου. Όταν όμως είσαι ένας διαφορετικός οργανισμός μπορεί να μην θέλεις να τα αποκαλύπτεις όλα αυτά ε, διότι υπονομεύουν τη λειτουργία σου. και άλλες φορές ε, ε, δεν μας ενδιαφέρει να μάθουμε για τα δεδομένα ή για τους δείκτες που είναι ρυθμισμένοι, αλλά είναι πιο ε, σημαντικό να μαθαίνουμε τη μεθοδολογία. Εν πάση περιπτώσει, για τις αγορές λιανικής, εγώ θα πρότεινα να δημοσιοποιούνται και τα δύο, και η μέθοδος και τα δεδομένα. Πρέπει να δούμε βέβαια και τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ε, αναλόγως να γίνεται δημοσίευση με λογικό τρόπο. Είμαι υπέρ και του friend licensing και της διαφάνειας της χρεώσεις και στα τέλη και να μην υπάρχει διασταυρωμένη ε, επιδότηση χορήγηση έως μη όφιλε στα CSD. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ε, αντίπαλα συστήματα για τις τρίτες χώρες. Εμείς προσπαθούμε και είμαστε πρωτοπόροι τώρα ε, ε για την ΑΙΟΣΚΟ να κάνουμε νομοθεσία και δεν μας ακολουθούν πάντα οι άλλοι. Ε, θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε κριτήρια για τη συγκριτική αξιολόγηση με βάση την ΑΙΟΣΚΟ και να υπάρχουν ισοδύναμα αντίστοιχα στις νομοθεσίες. Ενδεχομένως χρειαστεί να τα αναθεωρήσουμε όλα αυτά και βάση των όσων ρυθμίζει παγκοσμίω η ΑΙΟΣΚΟ. Το έχουμε κάνει και αλλού αυτό ας πούμε, στα λογιστικά πρότυπα και αλλού. Δεν είναι κανένα απολύτως καινούριο θέμα, ούτε νέα ιδέα που κατατίθεται εδώ. Για το ρόλο της ΕΣΜΑ, της ΕΑΚΑ, ως προς το κρίσιμο σημείο ε, για τα benchmark, τους δείκτες αξιολόγησης, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Ο Γκέι Μίτσελ προτείνει μια διατύπωση Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη στη συνεδρίαση των σχεδόν, το έχουμε συζητήσει ήδη. Αυτό που προτείνει ο Γκέι Μίτσελ για την αιτιολογική σκέψη είναι καλύτερο ε, από το άρθρο. Ενδεχομένως... Η ΕΣΜΑ έχει μια αντίληψη για το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και η Άσκο βέβαια και η ιστορική εμπειρία. Και όταν ισχύει κάτι σε ένα κράτος μέλος, μπορεί να θέλει να διατηρήσει αυτό την εποπτεία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο αυτό ή πιθανό Ο ε, ε, δείκτης αναφοράς λοιπόν θα πρέπει να υποχρεώσει εκείνους που πρέπει να ενεργούν να ενεργήσουν. Αλλά ποιος έχει αυτή την ε, αρμοδιότητα. Αν περάσουμε στο IBOR, στους διαχειριστές δικτών διατραπεζικού επιτοκίου δεν ξέρω αν σκόπιμο κάτι Το συζητούμε και θα συνεχίσουμε να το συζητούμε σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών. Θα πρέπει να βρούμε μια σωστή γραμμή που να μπορεί να λειτουργεί στην πράξη. Και τέλος, τα παραρτήματα δεν είχα ε, χρόνο να ασχοληθώ ε, με αυτά να το συζητήσουμε με τους σκιώδεις. Τι προτείνω εγώ, όσο γίνεται να γραμμιστούν με το ΑΙΟΣΚΟ, ε, να είναι αναλογική, ιδιαίτερα τα παραρτήματα 3 για τα εμπορεύματα για να λαμβάνουμε υπόψη ε, οποιαδήποτε νέα εξέλιξη, ακόμα και να αναβάλουμε τη θέση σε ισχύ σε, για χρόνο, όταν ξέρουμε ότι έχει ρυθμιστεί το θέμα της ΑΙΟΦΣΚΟ. Εγώ με χαρά να ακούσω τις προτάσεις σας για να το διατυπώσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρω ότι ορισμένοι βουλευτές θέλουν από τώρα πλήρη εξαίρεση ε, και κάποιοι άλλοι που δεν τους ικανοποιεί αυτή η πρόταση. Να οριστούν πρώτα ε, ε, τα κριτήρια αιώσκο και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τους και τώρα να μας πούν για τις τροπολογίες τους και τις απόψεις τους για το πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Γκέι Μίτσελ, κάπου τον είδα, εδώ είναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνήθω ε, κάνατε μια πολύ δίκαιη και πλήρη επισκόπηση. Με ενδιαφέρον άκουσα αυτά που κάνετε πάνω στο θέμα αυτό. Της ε, τροπολογίε μου τις έχω επικεντρώσει κυρίως ε, στον ρόλο της ΕΣΜΑ, τη ΕΑΚΑ και τίθεται πάλι το θέμα των κατακελώντων, των whistleblowers. Πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει επαρκής ε, ρύθμιση για το θέμα αυτό. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, θα ήθελα να επαναλάβω τη στήριξή μου προς ε, την προσέγγιση της εισηγήτριας. Είναι, πολύ... Είναι πολλές και διαφορετικές οι τροπολογίες ε, πάνω στο θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν προσεκτικά το θέμα του πεδίου εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε κατά νου τις αρχές της ΙΟΣΚΟ όταν το κάνουμε αυτό και να εφαρμόσουμε τον κανονισμό με τρόπο αναλογικό σε σχέση με τα χαρακτηριστικά, τα ευάλωτα σημεία και τους κινδύνους ε, των διαφόρων ε, benchmarks, κριτηρίων αξιολόγησης. Και ως προς την αιτιολογική σκέψη για την ΕΣΜΑ, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε εμείς οι σκιώδες συζητητές σε συνεργασία μαζί σας να βρούμε μια λύση. Οι τροπολογίες μου που λένε ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να μπορεί να αναθεωρεί κάποια benchmarks ε, εκτός ε, αν ε, στα κράτη-μέλη υπάρχει επαρκή σε ρύθμιση, μου φαίνεται ότι λειτουργεί καλά. Στις, υπό τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει η ΕΣΜΑ να αναθέτει τη δουλειά αυτή στις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές. Και το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά ε, χρήστες και ενδιαφερομένους σε πάνω από ένα κράτος μέλος, ε, το οποίο σημαίνει ότι η ρύθμιση ενός κράτους μέλους μπορεί να μην καλύψει επαρκώς τους κινδύνους αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος δεν έχει επαρκή εποπτεία, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε μία περίπτωση στα κράτη-μέλη μας όπου να μην ισχύει αυτό. Και όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά κάποια βασικά αγαθά, Βλέπω ότι έχουμε την τροπολογία 417 του Όλε Σμιτ. που τονίζει μια διαφορετική πτυχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να την εξετάσουμε αυτή με ανοιχτό πνεύμα. Ας ακούσουμε τι έχει να πει και ο Βέρνετ για την ε, εξαίρεση των ε, βασικών αγαθών ούτως ή άλλως. Όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας, πολλοί είπαν ότι τον επιβάλλουμε έναν τέτοιο κώδικα σε μικρούς ε, συνεισφέροντες, σε λιγότερο σημαντικούς, ε, δεν θα λειτουργήσει πολύ καλά στην πράξη. Σημειώνω ότι κάποιοι από εμάς ε, έχουν συμπεριλάβει διατύπωση που να κάνει πιο χαλαρή τη διάταξη για τον κώδικα δεοντολογίας. Κυρία Πρόεδρε, άλλοι από εμάς ζητάμε να είναι πιο δεσμευτικός ο κώδικας δεοντολογίας. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πιο σωστό. Και έτσι ο, ο κόσμος δεν θα υποβάλει ελαφρά την καρδία ε, σχετικές πληροφορίες. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν διαχωρισμό σε κατηγορίες ώστε για ε, τα κρίσιμα benchmarks να υπάρχει νομική δέσμευση ενώ για τα άλλα να υπάρχει πιο ε, χαλαρή προσέγγιση. Επίσης, ε, οι τροπολογίες μου ενσωματώνουν τις αρχές της ΙΟΣΚΟ που εξετάζουν τον κίνδυνο κατά τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης. Το επίπεδο διαφάνειας που απαιτείται θα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης στα στοιχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα ε, στα δεδομένα ανάλογα με το από πού προέρχονται. Και κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ νομίζω μαζί σας στο σημείο αυτό όσον αφορά τα κρίσιμα benchmarks Η μεθοδολογία για τον καθορισμό τους ε, θα πρέπει να εξαρτάται από τις ε, πηγές. Πιστεύω ότι είναι καλό αυτό το άρθρο να διαχωριστεί σε διάφορα μέρη και να είναι σαφές σε ποια δεδομένα θα ε, δημοσιεύονται σε ποια περίπτωση. Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, τα σχετικά άρθρα θα πρέπει να τα εξετάσουμε ιδιαίτερα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή δεν έχουν ε, αναλάβει βήματα για την εφαρμογή των αρχών της ΙΟΣΚΟ από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν είμαι βέβαιος αν ισχύει αυτό. Γίνονται πολλές συζητήσεις σχετικά με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην κλείσουμε τις αγορές μας απέναντι σε διαχειριστές από τρίτες χώρες. Ε, κυρία Πρόεδρε, εσείς και εγώ όμως έχουμε υποβάλει τροπολογία ώστε ένας διαχειριστής από τρίτες χώρες να ε, συμμορφώνεται με την ευρεία έννοια με τις αρχές της ΙΟΣΚΟ. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω την πρότασή μου για την ισοδυναμία, κάτι που αναφέρεται και σε άλλα νομοθετήματα. Αυτό μπορεί να ασκήσει πίεση σε τρίτες χώρες, να παράσχουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να βασίζεται στις αρχές της ΙΟΣΚΟ. Κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Και τέλος, Θέλω να επανέλθω στη σημασία να διασφαλίσουμε ένα σύστημα καταγγελόντων. Οι whistleblowers να μπορούν να ε, ε, αναφέρουν απευθείας ε, στην ΕΑΚΑ ή αλλού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αντιπίνων. Κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει ο καθένα μα να διαβουλευτεί με την πολιτική του ομάδα. Νομίζω όμω ότι με τον τρόπο που το έχουμε χειριστεί μέχρι στιγμή πλησιάζουμε ε, σε ένα στάδιο όπου μπορούμε να εξετάσουμε πιθανού συμβιβασμού. Θα υπάρξουν βέβαια και τομεί όπου δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, θα πρέπει να του αντιμετωπίσουμε. Σα ευχαριστώ για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. Και τώρα η Έμιλη από του σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η κατάσταση είναι σαφής με την έννοια ότι ξέρουμε ότι έχουμε πολλές τροπολογίες που πηγαίνουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ε, ε, μιλάμε για ορισμούς. Επίσης ε, υπάρχουν και κάποιοι ορισμοί οι οποίοι μας, προσωπικά μας δημιουργούν προβλήματα, major benchmarks κτλ. Ε, πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί με τους ορισμούς και αυτό με προβληματίζει για την ώρα. Κάτι άλλο. Οδηγούμαστε προς μια πιο περίπλοκη πρόταση από αυτήν της Επιτροπής και επίσης μια πρόταση που ίσως δεν έχει το εύρος της αρχικής προτάσεως της Επιτροπής. Ε, ακόμα και όσον αφορά την ίδια την ΕΣΜΑ, την ΕΑΚΑ. Αυτό και αυτό έχει προκύψει στις συζητήσεις μας μεταξύ σκιωδών, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Θα κάνω μερικά σχόλια ε, σε κάποια σημεία που τα θεωρώ κρίσιμα πεδίο εφαρμογής. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θέλουν να επιτύχουν έναν, ένα όσο γίνεται μεγαλύτερο πεδίο. Ε, οτιδήποτε δηλαδή ε, περιορίζει το πεδίο δεν μας βρίσκει σύμφωνος και αυτό το κατέστα σαφές. Επίσης είπατε από την αρχή ότι δεν θέλετε να εστιαστείτε πολύ στους διαχειριστές και αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό. Απ' την άλλη πλευρά ωστόσο, πρέπει να ε, βρεθούν ε, σαφείς απαιτήσει για τους παρόχους. Ε, γιατί υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας ο οποίος θα πρέπει να συνδεθεί με την κατάσταση και να είναι κατά κάποιο τρόπο πιο δεσμευτικός, αλλά ε, δεν λέω να είναι υποχρεωτικός ο κώδικας, αλλά να υπάρχουν κάποια ε, σαφώς καθορισμένα στοιχεία. Όσον αφορά το, ε, τους κρίσιμους δείκτες αναφοράς, critical benchmarks, θα πρέπει να είναι κρίσιμοι για το σύνολο της Ευρώπης και αυτό είναι λίγο προβληματικό. Επίσης θα πρέπει να βρούμε κάποιους ορισμούς που να ισχύουν όχι μόνο για τους ε, τώρα ισχύοντες μεγάλους δείκτες αναφοράς αλλά να είναι πιο μακρόπνοοι ε, και να είναι αρκετά κρίσιμοι έτσι ώστε να έχουν ε, και μακρά διάρκεια ζωής, ποιότητα και χρονική διάρκεια μεγάλη. Έτσι θα πρέπει να οριστούν οι κρίσιμοι δείκτες αναφοράς. Και επ' αυτού νομίζω θα πρέπει να δουλέψουμε. Όσον αφορά την ΕΣΜΑ ΕΑΚΑ, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θέλουν η ΕΣΜΑ να έχει ρόλο ε, σε, στα, στους κρίσιμους δείκτες αναφοράς, κρίσιμους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να κινείται όχι μονάχα ε, για τον ορισμό ε, ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, αλλά ε, να έχει και τη δυνατότητα παρέμβασης όταν μιλάμε για κρίσιμους δείκτες αναφοράς. Επίσης έχουμε κάποια σημεία, αν όχι αντίρρησης, αλλά συζήτησης επ' αυτού. Όσον αφορά τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, νομίζω ότι το θέμα είναι και ευαίσθητο και δύσκολο και θα ήθελα να πω σε όλους και στην Κομισιόν ότι οι σκέψεις ε, που κάνουν, δηλαδή να επιβάλλουν υποχρεώσεις ε, και στους ε, διαχειριστές τρίτων χωρών, είναι ενδιαφέρουσα σκέψη, αλλά θα πρέπει να δούμε, και το έχουμε συζητήσει και μεταξύ σκιωδών, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. υποχρεωτικές ε, ε, δεσμεύσεις για τους, ε, για τους διαχειριστές δικτών αναφοράς τρίτων χωρών είναι ένα ευαίσθητο θέμα και δεν νομίζω ότι εδώ αρκούν οι αρχές της ΙΟΣΚΟ, δεν είναι δεσμευτικές αυτές και διακινδυνεύουμε ε, απλώς η βιομηχανία παροχής δικτών αναφοράς να μετακινηθεί, να μετατοπιστεί εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα κύρια σημεία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας ε, σε αυτή τη θητεία. Ξέρω ότι και το Συμβούλιο δεν δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα, δεν προχωράει πολύ γρήγορα, αλλά τουλάχιστον εμείς το δικό μας κομμάτι με τους ορισμούς μας, τους σαφείς και τους καθαρούς, ε, γιατί να, την έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε δει τι έγινε και πέρσι με την χειραγώγηση δικτών αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Φιλίπ, καλημέρα σε όλους σας. Πολύ καλά κάνουμε και ασχολούμαστε με αυτό το σημαντικό θέμα, γιατί ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί. Το σκάνδαλο για τα ε, ε, για τα επιτόκια της Forex όσον αφορά το Libor ε, είναι πολύ μεγάλο και τώρα ξετυλίγεται σιγά σιγά. Μόλις άκουσα την φίλη και συνάδελφο Έμιλη, έχουμε μιλήσει μαζί. Ε, συμφωνώ μαζί της όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, πρέπει να είναι πρακτικό το πεδίο εφαρμογής και να μπορεί ε, να λάβει υπόψη ε, όλα τα στοιχεία και τις αντιρρήσεις κτλ. Ε, ξέρω Σάρων ότι δεν είσαι πολύ Βρετανική Βρετανής, είσαι πιο πολύ Ευρωπαία Βρετανής, μπορείς να το δουλέψεις αυτό λίγο. Στους, στη συνάντηση των σκιωδών είπαμε ότι θα πρέπει να περάσουμε, να, ξεπεράσουμε μάλλον τα καθαρά τεχνικά πρότυπα. Αυτό άλλωστε κάνουμε και για τις τράπεζες. Ε, να δούμε δηλαδή το δυνατό τη δυνατότητα εποπτείας όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς, θέλετε να τους ονομάσετε κρίσιμους, θέλετε να τους ονομάσετε κάπως αλλιώς, ε, εν πάση περιπτώσει για δείκτες αναφοράς οι οποίοι έχουν επίπτωση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η ΕΣΜΑ να είναι ε, δεσμευμένη. Υπάρχουν οι εθνικές αρχές ε, οι οποίες ε, ε, μπορούν ενδεχομένως με ανάθεση της ΕΣΜΑ να ε, ε, κάνουν ε, κάποια εποπτεία, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Ωστόσο, το θέμα της εποπτείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εποπτεία λοιπόν δικτών αναφοράς που μπορεί να έχει μεγάλη επίπτωση στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να είναι αυτή η εποπτεία αρμοδιότητα μιας αρχής. Εδώ βέβαια προκύπτει το ευαίσθητο ζήτημα το πώς θα μοιράσουμε την αρμοδιότητα μεταξύ αρμοδιότητα επιλογής και αρμοδιότητα εκτέλεσης. Ε, οι ορισμοί των διαφορετικών κατηγοριών δικτών αναφοράς, αυτό η ε, κατανομή είναι δύσκολη και περίπλοκη. Νομίζω ότι θα πρέπει απλώς να ορίσουμε κάποια ποσοτικά και ποιοτικά κατόφλια ανακατηγορία. Υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι απασχόλησε μόνο εμάς, είναι ε, το κατά πόσον είναι δόκιμοι οι, δείκτες, οι αναφοράς. Εξηγούμε οι δείκτες αναφοράς ε, ε, οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι αντίστοιχοι με, με τι. Δηλαδή γιατί χρησιμοποιούμε ε, τον Λίμπορ για την βιώσιμη εξέλιξη επιτοκίων στα ενυπόθηκα δάνεια ας πούμε. Αυτό εννοώ όταν οι δείκτες αναφοράς χρησιμοποιούνται για κάτι για το οποίο δεν είναι σωστά επιλεγμένοι, δημιουργούν στρεβλώσεις και κινδύνους. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί με κάποιο τρόπο. Μπορεί κανείς βεβαίως ορθώς να πει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο ε, στο οποίο μπορούμε σαφέστατα να καθορίσουμε ε, ποιο ε, είναι ο σωστός τρόπος χρήσης του συγκεκριμένου δείκτη αναφοράς και ενδεχομένως προχωράμε πολύ μακριά στον καθορισμό του ε, τι πρέπει να κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να καλέσουμε τουλάχιστον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα ε, τα επόμενα χρόνια και να υπάρχει βεβαίως και στην ρήτρα αναθεώρησης έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο ε, μη δόκιμης χρήσης των δικτών αναφοράς. Θα ήθελα και εγώ να υπάρχει όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια. Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα λέμε ότι θα πρέπει η διαχείριση των, των ε, εταιριών να γίνεται, να οδηγείται κατά κάποιο τρόπο από την αγορά. Εντάξει, λοιπόν, εμείς ζητάμε μεγάλη διαφάνεια στις αγορές και αυτοί που λένε ότι η υπερβολική διαφάνεια μπορεί να παρεμποδίσει ε, την σωστή λειτουργία των αγορών, εγώ λέω ότι αυτό θα πεφευχθεί αν η διαφάνεια των αγορών ε, ξεκινήσει από την αρχή. Ε, Επίσης, ε, όσον αφορά τα παραρτήματα και τις τροπολογίες, ακόμα δεν έχουμε δει ποια είναι η πρόθεση της ε, Σάρων, θα περιμένουμε και θα δούμε. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό είναι απόλυτα ικανοί και ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε σε κάτι ικανοποιητικό. Ευχαριστώ. Ποιος εκπροσωπεί τον Σαϊτ Κεμάλ? Στέισακ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Σκέφτης ηγητής μας είναι ο κύριος Ατζήτη Καμάλ ε, και με παρακάλεσε να σας παρουσιάσω μερικά από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του, διότι δυστυχώς έχει άλλη ανηλυμένη υποχρέωση και κολλιέται να παρευρεθεί. Είναι δύσκολο να τον αντικαθιστά κανείς, ε, όπως βλέπετε. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον εκπροσωπήσω. Χιούμορ έχεις λέει, πάντως λέει ο κύριος Λάμπραχτς. Μα Φίλιπ, γι' αυτό είσαι από τους πιο αγαπημένους μου πρασίνους εσύ. Ευχαριστεί την εισηγήτρια ο κύριος Καμάλ και τους Κιώδης για την ε, καρποφόρα συνεδρίαση του Στρασβούργου την περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται να υπάρχει ευρία συνένεση σχετικά με την ανάγκη να αποκρισταλωθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τις εκλογές του Μαΐου. Ο κύριος Καμά παραμένει ανησυχών για το πεδίο εφαρμογής ότι είναι υπερβολικά ευρύ ε, πιστεύει ο κύριος Καμάλ ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε τους δείκτες εκείνους αναφοράς που είναι ευάλωτοι για χειραγώγηση και προσφέρονται όπως είναι οι διάφοροι δείκτες IBOR ή ε, οι κρίσιμοι δείκτες αναφοράς που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και δεν θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα πάντα ως αυτοσκοπό. Αυτή είναι μία από τις βασικές θέσεις του κυρίου Καμάλ. Ο Σαΐντ και που προτείνουμε η εποπτεία του Λάιμπορ να παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπεται με τον κανονισμό αυτό και είναι πρωτοπόρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα πρέπει να υπονομεύουμε συστήματα που λειτουργούν ήδη σε κάποιο κράτος μέλος για την ΕΣΜΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών ε, και Αγορών, θα πρέπει να ρυθμίζει τις αρμόδιες αρχές, αλλά δεν πρέπει να την παραφορτώσουμε με περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες από τις οποίες μπορεί να αντέξει. Έγινε λόγος και για τον κώδικα δεοντολογίας, αν θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικός ή όχι. Ο κύριος Καμάλ δεν είναι πεπισμένος ότι θα πρέπει να είναι δεσμευτικός δεδομένου ότι αυτό θα καταλήξει σε ε, λιγότερες εταιρείες που αναφέρουν τα κριτήρια και τους δείκτες αναφοράς. Μας ενδιαφέρει η σωστή λειτουργία χωρίς να υπερβάλλουμε όμως. Δηλαδή να μην ρυθμίζουμε υπερβολικά κάποια πράγματα που κανείς δεν θα δηλώνει. Ε, περιμένει την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών για συγγνώμη των εισηγητών και περιμένει μια λύση που θα είναι και αναλογική και ευέλικτη. Και προσβλέπει βεβαίω και φυσικά στην περαιτέρω συνεργασία σα. Ευχαριστώ. Uh, uh, Έχω ένα κατάλογο μιλητών. Βέρνερ Λάγκερ, Σιλβί Γκουλάρ, άλλο κανεί θέλει να προσθέσουμε το όνομά του. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να σας κάνουν, αλλά μπορεί και όχι. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την στρατηγική της εισηγήτριας. Σε μισή ώρα ξεκινάει ψηφοφορία στην Επιτροπή Βιομηχανίας για τους δείχτες αναφοράς για τις πρώτες ύλες. Δεν μπορώ λοιπόν να σας αναφέρω ακόμα το αποτέλεσμα τις ψηφοφορίε για την έκθεση τη κυρία Ματία. Υπάρχουν πολλές τροπολογίε. Μου φαίνεται όμως απαραίτητο, πέρα από, τα, πέρα από τους οικονομικούς δείκτες αναφοράς, να ασχοληθούμε και με τους δείκτες για πρώτες ύλες που κυρίως βασίζονται σε δεδομένα από τρίτες χώρες που δεν ρυθμίζονται και γι' αυτό δεν είναι δυνατό να υπάρχει διαφάνεια. Αν αποκλείουμε συνεισφέροντες ή επιβάλλουμε υπερβολικές απαιτήσεις, ε, ε, τότε κάτι θα έχουμε κερδίσει και στις περιπτώσεις ε, όπου κάποια αγαθά αποτελούν τη βάση, οι περιπτώσεις αυτές είναι διαφορετικές από, την, από τον χρηματοοικονομικό τομέα διότι σε κάποιες περιπτώσεις εξαρτόμαστε, Μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να νομοθετούμε ε, πολύ επιφυλακτικά. Διότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν κρατικές εταιρείες ε, που δεσπόζουν στον τομέα και είναι δύσκολο να βελτιώσουμε την διαφάνεια και τη βάση για τους δείκτες αναφοράς. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, αλλά γνωρίζουμε ότι στα, στους δείκτες αναφοράς Πέρα από τους ε, διαχειριστές υπάρχουν ε, κάποιοι παρατηρητές, ε, κάποιοι συνεισφέροντες από τον ιδιωτικό τομέα και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε να μην περιορίσουμε τη θελοντική συνεισφορά στοιχείων και έτσι να γίνει πιο αδιαφανής η αγορά αυτά που υπόθηκαν για την χρηματοοικονομική αγορά. Νομίζω ότι μας βρίσκουν σύμφωνους και παρακαλώ την εισηγήτρια μετά την σημερινή ψηφοφορία στην Επιτροπή Βιομηχανίας να εξετάσουμε μαζί εάν μπορούμε να λάβουμε υπόψη τη θέση της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ε, ευχαριστώ για τα υπόλοιπα, με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ πολύ, Σιλβί. Ευχαριστώ, Σάρων. Ευχαριστώ όλους. Όπως είπε και ο Φιλίπ προηγουμένως, ε, η συγγήτρια ε, μάλλον και ε, Σκιώδης είναι πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ευρεία προσέγγιση, κυρίως ε, με τρόπο ώστε η Ευρώπη τελικά να μην βρεθεί... Ε, κάτω από το όριο ας πούμε των ε, ε, απαιτήσεων. Δηλαδή ε, με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους δείκτες αναφοράς ε, μπορούμε να φτάσουμε ε, σε ένα ευρύ πεδίο αποχρώσεων. Δεύτερον, πιστεύω ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι όχι μονάχα δικαστικού χαρακτήρα αλλά διοικητικές και ηθικές κατά κάποιο τρόπο. Ίσως αυτό εξαρτάται από τις διαφορετικές νοοτροπίες. Τροπολογία 23 η οποία πλέον μετά την χθεσινή η απόφαση του δικαστηρίου παίρνει άλλη απόχρωση. Ε, ε, ε, ξέρουμε ότι χθες έλαβε μια απόφαση στο δικαστήριο όσον αφορά το short selling και επομένως δίνει τη δυνατότητα στην ΕΣΜΑ, στην ΕΑΚΑ, να παίρνει συγκεκριμένες ακυρωτικές αποφάσεις και για τον ε, δίκτυ Λίμπορ και για άλλους ε, δίκτες που θα δει η συγγήτρια θα πρέπει να ε, πάρουμε κάποιες άλλες αποφάσεις. Οι αρχές πλέον όσον αφορά και την διαχείριση τύπου Μερώνη όπως είναι γνωστή αλλά και άλλες πλέον θα πρέπει να τις δούμε κάτω από ένα διαφορετικό φως. Ο Φιλίπ νομίζω ότι ε, θα πάρει τη θέση της ε, Πασκάλ και εν πάση περιπτώσει εγώ της έστειλα χθες ένα μικρό mail λαμβάνοντας υπόψη την χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου η οποία δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας. Πρόεδρος, ε, θέλει να... όχι, η Κομισιόν θα πάρει το λόγο, δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την συζήτηση που δείχνει ότι το Κοινοβούλιο πολύ σοβαρά ε, παίρνει την πρόταση αυτή που είναι σημαντική. Το θέμα των δικτών αναφοράς δεν συζητείται μονάχα στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. και βεβαίως ακόμα περισσότερο ε, στις, ε, στην ΑΙΟΣΚΟ που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των αγορών. Θα ήθελα ε, να πω ότι η πρόταση της Κομισιόν σκοπό έχει να τεκμηριώσει την ακεραιότητα των δικτών αναφοράς. Θεωρήσαμε ότι ότι η έλλειψη σύγκρουσης ε, συμφερόντων, η καλή ε, και ταυτισμένη μεθοδολογία, η διαφάνεια είναι στοιχεία ε, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη στην παροχή δικτών αναφοράς και βεβαίως να ακολουθούνται και από άλλα παρεπίμπτοντα όπως ας πούμε η δήλωση, η κοινοποίηση του υπεύθυνου παρόχου. Όσον αφορά το πεδίο αναφοράς, ε, εφαρμογή, συγγνώμη, πρέπει να πω ότι βασιστήκαμε στα πρότυπα ε, της ΙΟΣΚΟ, τα οποία έχουν ευρύ πεδίο και αυτό γίνεται με τρόπον ώστε οι διαφορετικές αξιολογήσεις και τρόποι αναφοράς, ε, ανατομέα δικτών αναφοράς, έχει προκύψει ότι όλοι αυτοί οι δείκτες αναφοράς, λέω, ε, έχουν τροτά σημεία και επομένως ε, πρέπει να διασφαλίσουμε το, το σωστό επίπεδο ρύθμισης ε, και βεβαίως όσον αφορά τα παράγωγα ε, των, ε, και όσον αφορά τις, τις παράγωγες αγορές δηλαδή των βασικών αγαθών και εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα πρότυπα ΙΟΣΚΟ διότι η ΙΟΣΚΟ έχει συγκεκριμένους τρόπους για την μεθοδολογία αναφοράς ε, επίσης στην Ιόσκο δεν υπάρχει δυνατότητα camp out για, τη, για τα παράγωγα και για τα ε, βασικά εμπορεύματα και για τα παράγωγα. Όσον αφορά την ΕΣΜΑ, εποπτικό ρόλο και επιπλέον συμπληρωματικούς ρόλους, πρέπει να πω ότι η Κομισιόν καλοδέχεται την, ε, τις γενικότερες ε, σκέψεις που ακούστηκαν εδώ, ε, διότι θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν αργότερα και συγκεκριμένες ρήτρες όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις. Πρέπει να πω όμως ότι η Κομισιόν στην πρότασή της το θέμα της εποπτείας των διαχειριστών δικτών, αναφοράς δίνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Θεωρούμε ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι παίχτες διότι γνωρίζουν καλύτερα την αγορά και θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν ο πλέον δόκιμος τρόπος. Ε, ωστόσο ε, το κολέγιο των ε, επιβλεπόντων μπορεί και των επιτηρητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να, γίνει μάλλον με κολεγίου ενεργειακό τρόπο. Τρίτες χώρες. Κατά την άποψη της Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να, υπάρχουν, να υπάρχει ισοδύναμο σύστημα στην πρόταση αυτή, γιατί όπως υπόθηκε άλλωστε, το να είμαστε η πρώτη στα πλαίσια των G20 που να κάνουμε τέτοια νομοθεσία θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, μία κατάσταση κατά την οποία όλοι οι υπάροχοι δικτών αναφοράς ε, θα πήγαιναν εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως έτσι ώστε να βρουν ε, ευνοϊκότερους και λιγότερο αυστηρούς όρους. Δεν θέλουμε να κλείσουμε λοιπόν την ευρωπαϊκή αγορά, επομένως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δείκτες αναφοράς ε, παρέχονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με, αντίστοιχα, με αντίστοιχους όρους ε, με ό,τι ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δείκτες αναφοράς για τη συνεγκρισιμότητα είναι τα πρότυπα της ΙΟΣΚΟ για την χρηματοπιστωτική συγκρισιμότητα. Ε, υπάρχει δυνατότητα βεβαίως επιπλέον ευελιξίας όσον αφορά την αξιολόγηση ισοδυνάμων, όσον αφορά το ερώτημα το κατά πόσο είναι σημαντικό ή όχι ε, αυτοί οι πάροχοι δικτών σε τρίτων χωρών να εποπτεύονται από ρυθμιστές, θεωρούμε ότι αυτό είναι ουσιώδου σημασίας, απόλυτα ουσιώδου σημασίας. Το γεγονός ε, ότι ε, ε, ε, κάποιος πιστοποιεί συμμόρφωση με τους κανόνες είναι απαραίτητο γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπήρχε έτσι μία ίση αντιμετώπιση όλων των παρόχων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα σύντομα μόνο να συνοψίσω. In the, uh, compromises στις συμβαστικές προτάσεις που έχουμε υποβάλει υπάρχουν κάποια άρθρα που όντως θα χρειαστεί ε, κάποια υποπαράγραφος για να υπάρξει διαφορετική ταξινόμηση σε κατηγορίες. Ας πούμε, πώς αντιμετωπίζονται οι ε, συνεισφέροντες σε σχέση με αυτά που είπε ο Σαΐτ Καμάλη. Είναι τεράστιο το φάσμα. Ορισμένοι περίπου αυτόματα εισάγουν αυτές τις πληροφορίες πάρα πολύ συχνά, για να μην πω και σε πραγματικό χρόνο. Και πολλά είναι σε θέλουσια βάση. Και αν τρομάξουμε πάρα πολύ τον κόσμο δεν θα δηλώνει τίποτα. Και δεν θα έχουμε και τους δείκτες και τα κριτήρια φοράς μας. Από την άλλη, όταν είναι αρκετά υποκειμενικό και κρίσιμοι δείκτες και σημαντικοί, χρειαζόμαστε έτσι πιο στεναρή αντιμετώπιση και πιο δυναμική. Θα πρέπει να τα μελετήσουμε όλα αυτά και θα σημειώσω τις διάφορες κατηγορίες που πρέπει να δημιουργήσουμε και θα αναδύονται παντού. Συμφωνώ με την Έμιλη ότι θα πρέπει να είναι απλό το πεδίο εφαρμογή, αλλά οι δείκτε αναφοράς είναι τόσο περίπλοκοι που θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζονται και διαφορετική μεταχείριση. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μπει σε μια γενική κατηγορία. Ξέρουμε ότι η ΕΑΚΑ έχει αρμοδιότητες ε, τις οποίες ασκεί και ε, εκτελεί σε πολλές περιπτώσεις ε, μια εθνική αρχή, ε, παρόλο είναι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό ε, στην ΕΣΜΑ για να διεκπαιρεώνουν όλες αυτές τις εργασίες. Χρειάζονται λοιπόν πραγματογνώμονες και εμπειρογνώμονες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για να κάνουν και μια εργασία έτσι, επιλογή στο τι έχει δηλωθεί και τι όχι, τι ισχύει και τι όχι. και να ανταποκρινόμαστε και στι αλλαγέ. Δηλαδή κάτι που δεν είναι κρίσιμο όσο δείξει αφορά σήμερα, μπορεί κάποια στιγμή να καταστεί. Εντάξει, να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω τι εννοούμε. Ε, τις ποιοτικές διαφορές δηλαδή των κρισίμων δικτύων, ε, δικτών συγγνώμη, αναφοράς. και χρειαζόμαστε και κάποιες προτάσεις Όλες οι εποπτικές αρχές το ζητούν από εμά για την ομοθεσία. Καταλαβαίνω αυτά που είπες εσύ Φιλίπ, δεν ξέρω. Αν έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου 100% ε, για το βασικό κίνδυνο ή το, το θεμητό ή το σκόπιμο. Δεν ξέρω για τους ε, ορισμούς αυτούς να το ξανακοιτάξουμε, να δούμε το περιτύλιγμα θέλετε. Γιατί κάποια στιγμή ε, μπαίνει και μύφιντ εκεί. Αν είναι σκόπιμη μια επένδυση ας πούμε ε, για το λιανικό καταναλωτή και τα λοιπά. Αν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμιά ιδέα γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη. Mm. Και θα μας βοηθούσε. Θα δούμε τι θα πει και η Επιτροπή Βιομηχανίας, θα το εξετάσω με ενδιαφέρον. Είχαμε προβλήματα με το MIFID γιατί δεν είναι στο REMIT. Και η λύση θα ήταν ενδεχομένως κάποια στιγμή να ενταχθούν και στο REMIT. Ε, αυτό πρέπει να το κάνει η Γενική Διεύθυνση ε, Αγορών, ΜΑΤ αλλά να τα έχουμε υπόψη μας για πιο μακροπρόθεσμη λύση σε πολλούς τομείς. Για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι για λόγους κατάχρησης αγοράς. Τα έχουμε ρυθμίσει πάρα πολύ καλά και πολύ προσεκτικά σε αυτή την νομοθεσία για να καλύψουμε και τα κριτήρια και δείκτες αναφοράς, γιατί θεωρήθηκε αδυναμία αυτό. Η Κατά λάθο ε, ήταν αδυναμία σε προηγούμενη νομοθεσία για να μην ξαναδούμε ή να μην επαναδιατυπώσουμε ε, την νομοθεσία για την κατάχρηση αγοράς θα πρέπει να παραπέμψουμε εκεί και να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο κάθε φορά καθεστώς επιβολής κυρώσεων. Ένα τελευταίο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δέχομαι ότι σε μερικές περιπτώσεις συμφωνείτε με την ΙΟΣΚΟ ενώ σε κάποιες άλλες όχι. Προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε την κατάσταση πολύ από εμά για τα προβληματικά σημεία. Ε, κάπου που έχει ε, διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η τιμολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων pricing instruments, αλλά καμία φορά είναι pricing assets, στοιχεία ενεργητικού. Δεν είναι πάντα ταυτόσιμο αυτό. Γι' αυτό αναφέρομαι στην EIS. Με χαρά να ε, μου εξηγήσετε η δική περί τίνος πρόκειται. Αλλά εγώ θέλω να αναφερόμαστε σε financial assets και σε financial instruments. Γιατί δεν ταυτίζονται πάντα αυτά τα δύο συνοψίζοντας ε, οδεύουμε προς μία λογική μάλλον προσέγγιση πιστεύω ξέρω ότι δεν θα ικανοποιηθούν οι πάντες αλλά πιστεύω ότι έχουμε πολλά κοινά και θα μπορέσουμε κάπου να τα βρούμε εν πάση περιπτώσει έτσι όλοι να είμαστε σχετικά ευχαριστημένοι ε, πάντα στα πλαίσια του Ιώσκο και να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα συμπεριλάβουμε όπως προχωρούμε, ε, όπως κάναμε και με τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Χρονοδιάγραμμα. Είπαμε. Θα αλλάξουμε την ψηφοφορία. Θα πάει στις 17 Φεβρουαρίου το αργότερο. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο χρονοδιάγραμμα και αν συμφωνείτε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε συγκεκριμένο για το Συμβούλιο ένα κείμενο για να μπορεί ε, να το εξετάσει όταν αρχίσει να συζητάει το θέμα και μπορεί και να τους ενθαρρύνουμε ε, όταν θα έχουμε δική μας πρόταση, να πούμε κοιτάξτε τι αποφασίσαμε εμείς ε, και να προωθηθεί τον Απρίλιο και μπορεί και να ανασκουμποθεί το Συμβούλιο, ποιος ξέρει, για να τα βρούμε. Εμείς το, το προσφέρουμε ως κίνητρο, ως καροτάκι. Αυτά. Ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα στο θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης. που είναι η έκθεση συνεκτικότητας. Ε, λάβαμε κάποιες τροπολογίες από τους συντονιστές, διότι νομίζω ότι Από τεχνικής πλευράς είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε πολλούς ε, σκιώδεις. Θα σας πω ποια είναι η κατάσταση και όποιος άλλος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίσα Φερέιρα και τον Μπέρχαρτ ε, Πάλς για τις επικοδομητικές τροπολογίες τους ε, για την έκθεση σχετικά με την συνεκτικότητα της νομοθεσίας για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή τώρα που πλησιάζει στο τέλος της η θητεία μας για να βοηθήσουμε τους συναδέρφους στην επόμενη θητεία. Αποτελεί και εξέταση του τρόπου που έχουμε εργαστεί σε αυτό το τομέα πολιτικής. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε ευρεία ε, διαβούλευση με διάφορε ομάδε ενδιαφερομένων που πραγματοποιήθηκε το 2013 σχετικά με το πώ μπορεί να βελτιωθεί η συνεκτικότητα της νομοθεσίας ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τις υπηρεσίε. υπηρεσίες. Επικεντρωθήκαμε στην σχέση μεταξύ των διαφόρων νομοθετημάτων και τις διαδικασίες στα θεσμικά όργανα. Στην έκθεση αυτή κάνουμε κάποιες επικοδομητικέ προτάσεις προς τους διαδόχους μας και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ πώς ε, μπορούν να εξετάζουν ε, την ε, εφαρμογή νομοθεσίας που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο συχνά δημόσιες διαβουλεύσεις για να λαμβάνει συνεισφορές από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. Και Επίσης θα πρέπει η Επιτροπή μας να εξετάζει και την επιλογή των εισηγητών και σκιωδών. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, φτιάξει ένα ενιαίο νομικά δεσμευτικό μέσο για τις οικονομικές αγορές. Ε, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται οι μελέτες αντικτύπου και να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής. Επίσης ε, θα πρέπει να γίνονται συνδυασμένες αναθεωρήσεις των νομοθετημάτων που σχετίζονται μεταξύ τους. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή ανθρώπων εκτός της Επιτροπής ε, και Εάν κοιτάξουμε μία-μία τις ε, τροπολογίες, ε, η πρώτη εξετάζει την διαφορετική προσέγγιση παρόμοιων δραστηριοτήτων. Ε, η τροπολογία 2 για την παράγραφο 9 αναγνωρίζει ότι η Κομισιόν ε, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της ε, προσπαθεί να, ε, να καθιερώσει χρονοδιαγράμματα για την νέα νομοθεσία και αυτό αποτελεί χρήσιμη προσθήκη στην έκθεση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καλέσουμε τους συνομοθέτες να συνεχίσουν να παρέχουν βεβαιότητα στους ενδιαφερομένους όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα και πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα με την τροπολογία 5 του Μπέρχαρτ που τονίζει τη σημασία του να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων ε, χρηματοοικονομικών τομέων. Επίσης, ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας. Ε, κατά τον συνδυασμό των διαφόρων μαθητημάτων σε ένα ενιαίο νομικά δεσμευτικό μέσο. Δέχομαι ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν, αλλά αρκεί να δείτε την διολίστηση που είχαμε σε κάποιε από τι περιπτώσει νομοθετημάτων τη ε, χρηματοοικονομική αγορά, ε, ιδιαίτερα την, την έκθεση Λίκανεν που βρίσκεται ακόμα στην Επιτροπή και θα δημοσιευτεί σε ένα χρόνο όπου θα είναι πια τελείως άχρηστη και δεν ε, θα μπορέσει να λάβει υπόψη της την εμπειρογνωμοσύνη του παρόντος κοινοβουλίου. Η τροπολογία 3 για την παραγραφή 11 δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Εισάγει την πρόταση ε, ότι μπορεί να μην ε, είναι τόσο επιθυμητός ο συγκεκριμένος τρόπος επιλογής ε, των, των εισηγητών. Πιστεύω ότι σίγουρα ο τρόπος αυτός επιλογής θα συμβάλλει στην καλύτερη σχέση μεταξύ των διαφόρων νομοθετημάτων. Είμαι βέβαιη ότι στις μεγάλες πολιτικές ομάδες ε, τα μέλη θα θέλουν να νιώθουν ότι τους ανήκει. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάποιο είδους συγκέντρωση, κάποια είδους ομαδικής εργασίας. Ενδεχομένως να μπορέσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Στις μικρές πολιτικές ομάδες υπάρχει περισσότερη τάση συνεργασία επειδή υπάρχει ε, επικέντρωση στην τραπεζική πτυχή ή άλλες, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι θα είναι χρήσιμο αυτό και συχνά νιώθω ότι είμαι η αλλε αλλα δεν μπορουμε να αρνηθουμε οτι θα ειναι χρησιμο αυτο και συχνα νιωθω οτι ειμαι η μονη που έχω την ε, πλήρη εικόνα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια τριμερών διαλόγων. Αυτό είναι κάπως τρομακτικό. Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι. Επίσης δυσκολεύομαι να δεχτώ την τροπολογία 4 για την παράγραφο 14 καθότι αμφισβητεί την λέξη συνεκτικότητα όταν μιλάμε για τη σχέση ανάμεσα στους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς ε, που θεσπίζονται από άλλες δικαιοδοσίες. Βέβαια κάθε δικαιοδοσία είναι κυρίαρχη και μπορεί να αποφασίσει τους δικούς της ε, κανόνες, αλλά δεδομένης της ε, διασύνδεσης του παγκοσμίου χρηματοοικονομικού συστήματος, ένας τέτοιος συντονισμός είναι πολύ επιθυμητός. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς η νομοθεσία μας αλληλεπιδρά με κανόνες άλλων δικαιοδοσιών. Ε, και για, προτού να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις τους, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ε, ότι πέρα από τις ε, δικές μας συζητήσεις σε επιτροπή υποεπιτροπή της ΕΚΟΝ, η σύντομη αυτή έκθεση είναι πολύ χρήσιμη για να αποτελέσει σημείο αναφοράς και προσανατολισμό ε, στο Κοινοβούλιο που θα αναλάβει κατά την επόμενη θητεία. Επίσης ε, θα ήθελα το Κοινοβούλιο να σημειώσει τις παρατηρήσεις και συστάσεις στην έκθεση αυτή. Υπάρχει κανένα συνάδελφος που να θέλει να πάρει το λόγο. Αυτοί που έχουν υποβάλει τροπολογίες δεν είναι παρόντες. Mm. Δεν υπάρχει κανείς που θέλει να πάρει το λόγο. Ωραία. είναι κάτι το οποίο θα ψηφίσουμε κάποια στιγμή. 30 του μήνα νομίζω. Όπως σας είπα είναι έκθεση επιτροπής, δεν θα υποβληθεί στην Ολομέλεια. Είναι απλά ένας τρόπος ε, να μοιραστούμε κάποιες καλές πρακτικές. Με την βοήθεια της γραμματείας θα επικαιροποιήσουμε την έκθεση και θα την διανύμουμε εν ευθέτω χρόνο. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Η συγητής είναι ο Σαΐντ κατράουι. Είναι παρόν? Α, μάλιστα. Εξέταση των τροπολογιών. Έχει το λόγο, Σαΐντ. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι έχουν κατατεθεί παρακαλώ 433 τροπολογίες. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτή η έκθεση. Το έχω πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Θεωρώ ότι την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολύ καλή βάση για να εργαστούμε επί αυτής. Είναι ένα πρώτο συγκεκριμένο θέμα και φάκελος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων για να αντιμετωπίσουμε την παρατραπεζική ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω ένα υποκεφάλαιο που δεν είναι ίσως το πιο απειλητικό ή το πιο επικίνδυνο, αλλά καλό είναι να ρυθμιστεί σωστά. Για μένα τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ε, ε, θα πρέπει να διαδραματίζουν το ρόλο τους, δεν θέλουμε να το αποτρέψουμε. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ρευστότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια και η συμμεταχείριση όλων των επενδυτών. Πολλές από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή και μπορώ να τις υποστηρίξω. Εχθές συναντηθήκαμε με τους κοιόδους ηγητές και είχαμε μια πρώτη πολύ καλή συζήτηση πρέπει να πω και από ό,τι φαίνεται Υπάρχει ευρεία αντίληψη για μια σειρά σημείων, ιδιαίτερα για τη διεύρυνση ορισμένων προϋποθέσεων ε, για στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια, να επιτραπούν, να και τα ρέπος με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια και όρους. Ε, να μπορούν να ζητούν μια εξωτερική αξιολόγηση, stress test και να αναφέρουν ε, όλα αυτά βελτιώνουν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα κληθούμε να διευκρινίσουμε τις ερχόμενες εβδομάδες, τον τρόπο με τον οποίο ε, υπάρχουν ε, κάποιες απαιτήσει ρευστότητα και κεφαλαιακές πώς μπορούν να χαλαρώσουν λίγο ή να αυστηροποιηθούν οι κανόνες. Αυτό δεν το έχουμε λυμμένο ακόμα, το συζητάμε. Και τελικά θα πρέπει να σταθμίσουμε διάφορα πράγματα απέναντι και στην πραγματική οικονομία, αλλά να φροντίσουμε τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια να έχουν αρκετή ρευστότητα και να μην καταρρεύσουν. Και να υπάρχει δυνατότητα να επενδύουν, ας πούμε, σε ένα κεφάλαιο αμοιβαίων κεφαλαίων και θα πρέπει να διευκρινιστεί έτσι περαιτέρω ο ρόλος της ΕΣΜΑ, της ΑΚΑ. Το πιο κρίσιμο σημείο και επίμαχο είναι τι κάνουμε με τα περίφημα σύννευση και σχέση με τα λεγόμενα ε, Έχουν κάνει ε, κάποιες προτάσεις οι συνάδελφοι και τροπολογίες. Ε, πρώτη μου εντύπωση εμένα και θέση είναι να υποστηρίξουμε όσο γίνεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι έχει προτείνει ένα buffer η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα μαξιλαράκι εκεί. Ε, μια τριετία νομίζω. Εμείς θέλουμε μικρότερο χρονικό διάστημα, δηλαδή πιο γρήγορα να έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και μετά ε, από συστάσεις των διαφόρων εποπτικών αρχών ε, ευρωπαϊκών και παγκοσμίων προτείνουν να προ... Ε, χωρίσουμε προς τα φύνευση. Μια μελέτη του Χάρβαρτ ε, μιλάει, το Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε για 3-4% ως μαξιλαράκι. Βλέπετε αυτή είναι μια συζήτηση που δεν γίνεται ε, μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Οι αρμόδιες αρχές FSB και RSB προτείνουν να ξεφύγουμε από το ΣΥΝΑΦ και να περάσουμε στο ΒΙΝΑΦ. αυτού του είδους τα ταμεία ε, είναι δύσκολο να υποστηριχθούν όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Υπάρχουν προβλήματα ρευστότητα, αλλά τα σύναυσα έχουν μια ε, ιδιότητα χαρακτηριστικά που ε, εξασφαλίζουν οι επενδυτές σε περίοδους κρίσης να έχουν πλεονεκτήματα τύπου first mover. Λοιπόν, να αυξηθεί η ρευστότητα, η διαφάνεια. Ξέρω ότι ο κλάδος έχει τα δικά του συμφέροντα και δυσανασχετεί με μερικά από αυτά που προτείνουμε εμείς, αλλά τι να κάνουμε. Επίσης γίνεται λόγος για το λεγόμενο Fair Value Accounting. Δηλαδή, ε, πώς θα ε, καλύπτεται το κόστος και θα αποσβαίνεται το κόστος, ε, το ρίσκο και η ανάληψη κινδύνου. Ε, ε, υπάρχει διαφορά προφανώς στα αμοιβαία κεφάλαια σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις. Για τα σύναυση, οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές 10 με 15 ποσοστιαίες βασικές μονάδες ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και αυτό δεν συνάδει με την πραγματική αξία ε, των στοιχείων ενεργητικού. <laughs> Λοιπόν, ε, συνοψίζω και συμπεραίνω ότι ήρθε ο κύριος Δράγκη εδώ που μίλησε και υποστήριξε τη μετάβαση προς τα μεταβλητά αυτά κεφάλαια. Έχω πολλές ε, προτάσεις ε, να κάνω, είναι και πολλές οι θα τα συζητήσουμε. Εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία να περάσουμε στα βίνα τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτά τα buffers, τα μαξιλαράκια, να τα ενισχύσουμε, να τα συνδυάσουμε με μηχανισμούς ε, ρευστότητας και πιο περίπλοκα πράγματα. Είναι ένα εγχείρημα και μια άσκηση αρκετά ειδική. Λοιπόν, με χαρά περιμένω να ακούσω τις αντιδράσεις των συναδέλφων και σας ευχαριστώ ε, εκ των προτέρων για την επικοδομητική και καλή συνεργασία που έχω. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ, Σαΐντ. Ο Ζωάν Πολυγκοζές από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, ε, εισηγητή. Δεν το κάνω επειδή ήθιστε, το κάνω με μεγάλη ειλικρίνεια ε, γιατί πραγματικά η εργασία του είναι αποτέλεσμα κοινή εργασίας και σκέψης που μπορεί να μην έχει δώσει ακόμα συγκεκριμένα αποτελέσματα, ωστόσο η προσπάθεια εξέβρεσης συμβιβαστικών λύσεων είναι σαφής. Εδώ προσπαθούμε να ε, συνδυάσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια ε, ενώ ταυτοχρόνως θα συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση της πραγματικής ε, οικονομίας μέσω εργαλείων που είναι απαραίτητα γι' αυτό. Ε, επί των σημείων που η συγητής ανέφερε μόλις έχει εξευρεθεί ε, συμβιβαστική λύση έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται επενδύσεις ε, σε, άλλα, σε άλλα ομόλογα με όρους ασφαλείας. Άλλα σημεία τα οποία συζητιούνται ακόμα αφορούν τα θέματα της ρευστότητας ή της διαφοροποίησης παραμένει βεβαίως το ακαθόδες ε, ζήτημα των, των και των ΒΙΚΑΒ. Ε, δεν έχουν ταυτιστεί ακόμα, δεν έχουν καν προσεγγίσει οι απόψεις. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την συνεργασία μας είτε βάσει της προτάσεως της Κομισιόν είτε βάσει των προτινόμενων από τον εισηγητή γνωρίζοντας ότι αρκετοί συνάδελφοι επιθυμούν να μην ε, ε, διακινδυνεύσουμε ε, την κατάσταση των συνάψεων με στοιχεία τα οποία κατά τη βιομηχανία είναι απολύτως ουτοπικά. Έχουμε ξεκινήσει καλά και είμαι θετικά προσκύμενος προς την εργασία του εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ για την Άλντε όπως ε, λέει ο κύριος Κλίντσα, όπως είπε και ε, ο Σάνσφος Γκοζές, είχαμε πάρα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και συζήτησης. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις ε, πρώτες συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες μας υπέβαλε και τις οποίες μπορέσαμε να συζητήσουμε χθες το πιο ακαθόδες, μάλλον τα πιο ακαθόδη ζητήματα ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί, ως το άλλωστε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά σε μια συνένεση και επ' αυτών των θεμάτων. Μερικά σχόλια. Όπως ε, υπόθηκε και προηγουμένως, ο κύριος στόχος είναι να διασφαλίσουμε σταθερή ε, κατάσταση και ικανοποιητική ρευστότητα για να ε, μειωθεί ο κίνδυνος των λεγόμενων runs και ε, σε περίπτωση run, εν πάση περιπτώσει, να ε, υπάρξουν ήδη προαποφασισμένα μέτρα τα οποία μπορούν να εκτελεστούν άμεσα. Τώρα βεβαίως τώρα εάν θα είναι 20-25% τα ρευστά the quality of the assets of the basic Τα στοιχεία ενεργητικού ε, δεν μας απασχολεί τόσο πολύ, θα το βρούμε το σημείο αυτό. Ε, τώρα, όσον αφορά τα βίναυς με τα ε, υπέρ ή κατά, δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Ε, θα πρέπει να περάσουμε από τη μία κατηγορία στην άλλη οπωσδήποτε. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε να ε, ε, βελτιώσουμε τη υγεία των σύναψ και, και μέσα από τα ε, στοιχεία ανάνυψης τα οποία θα, και εξυγίανσης τα οποία τελικά θα επιλέξουμε. Νομίζω ότι όταν υπάρχει η δυνατότητα, όταν μάλλον υπάρχει το ενδεχόμενο ιδιαίτερα υψηλού και ανησυχητικού βαθμού εξηγιάνσεων να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί εάν ε, καταργήσουμε τα σύναψη και, τα υποχρεωτικά γίνουν όλα δύναψη, τότε ε, ε, αφαιρούμε μια δυνατότητα επιπλέον ρευστότητας που κάπου θα καταλήξει φαντάζομαι σε αποταμίευση στις τράπεζες, σε καταθέσεις ε, στις τράπεζες. Αλλά ε, μιλάμε όχι για εκατομμύρια, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά. Και νομίζω ότι θα αυξηθεί η αβεβαιότητα και η κίνδυνη των αγορών παντού. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Όσον αφορά το cost accounting, νομίζω ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το εισάγουμε, αλλά με προϋποθέσεις ε, σωστής, σωστού ελέγχου και ε, επιθεώρησης. Επίσης ε, υπάρχουν διάφορες συμβαστικές ιδέες οι οποίες έχουν ακουστεί και νομίζω ότι τελικά θα επιτύχουμε την τελική συνένεση. Ε, επίσης, οι κανόνες διαφοροποίησης. Σημαντικό. Θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε συγκέντρωση κινδύνων. Αυτό είναι πολύ, συγκεκριμένο, πολύ σημαντικό. Τελευταίο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι περιορίζουμε ή ακόμα και αποκλείουμε οποιαδήποτε ε, εξωτερική ε, βοήθεια ακόμα και κρατική ή οτιδήποτε. Είδαμε στο παρελθόν ε, πώς είχαν τα πράγματα. Ε, το, τα fans δεν το λένε βέβαια, αλλά ξέρουμε βλέποντας και τα στοιχεία ότι στο παρελθόν ε, υπήρχε τέτοια εξωτερική βοήθεια, ένα είδος sponsorship. Λοιπόν, είμαστε καθοδόν, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο μας. Οπωσδήποτε λοιπόν θα έχουμε ε, περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από τους πράσινους ο Φίλιπ Λαμπέρτσε. Γεια σας και πάλι. Καλημέρα Σαΐτ. Στα φλαμανδικά. Ναι, ναι. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ ε, ε, για το έργο του εισηγητού αλλά και για τις διαδικασίες ε, διαπραγμάτευσης. Εγώ θα συνεχίσω στα αγγλικά, γιατί στα αγγλικά τα έχω γραμμένα, έκανε την προσπάθεια αυτή, μίλησα μέχρι εδώ ολλανδικά, αλλά φτάνει. Πρώτη κρίσιμη ερώτηση. Ξεκινώ με την πιο σημαντική. Συνεχίζουμε να θέλουμε τα ΣΥΝΑΦ ε, στην ε, Ευρώπη, τις σταθερές ΚΑΕ. Ξέρω ότι η άκρα αριστερά ήθελε κατάργηση αυτών ε, των κεφαλαίων. Και μάλλον έχουν κάποιους λόγους ε, να υποβάλουν τέτοια πρόταση. Μερικές φορές είναι πολιτιστικά δύσκολα για δυτικοευρωπαίους να απαγορεύουν κάτι από το 1968 και μετά. απαγορεύεται η απαγόρευση. Αλλά εάν κάτι είναι κακό για την κοινωνία, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε την ε, απαγόρευση. Η ομάδα μας δεν είναι διαρρεμένη, ίσως επειδή είναι μικρότερη, αλλά δώστε μας μια ευκαιρία να γίνουμε μεγαλύτεροι για να δούμε αν θα παραμείνουμε ενωμένοι. Θα ήθελα λοιπόν ε, να καλέσω όλε τι άλλε πολιτικέ ομάδε ε, να μειώσουν εθελοντικά το δικό του μέγεθο ε, για να μεγαλώσουμε εμεί και να δούμε αν πράγματι θα μείνουμε ενωμένοι. Ε, πάντως εμείς είμαστε υπέρ της υποχρεωτικής μετατροπής των ΣΥΝΑΒ σε ΒΙΝΑΒ, σε ε, ε, κειμενόμενες καθαρές αξίες ενεργητικού, με κάποιο μεταβατικό διάστημα. Εάν... Ε, θέλουμε επίσης αυτές οι προϋποθέσεις ε, να ε, εφαρμοστούν μόνιμα. Επίσης θέλουμε κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις στη μεταπατική περίοδο. Καταρχάς, να υπάρχει αποθεματικό ασφαλείας, το NAV buffer δηλαδή, και ξέρουμε ότι ο Ζων Πολ έχει προτείνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης ε, να έχουμε αποθεματικό ασφαλείας αντισυγκυριακό. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια πρόταση αποκλειστικά δική μας. Ε, θα πρέπει να γεμίζεται το αποθεματικό αυτό όποτε υπάρχει θετική διαφορά. Πρόκειται για μη συμμετρική προσέγγιση στο buffering στα αποθεματικά αυτά. Επίσης ε, τα ΣΥΝΑΦ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί ε, η αξία των ε, στοιχείων του ενεργητικού. Νομίζω ότι αυτό το πρότεινε Σαΐντε στην τροπολογία 24. Επίσης να υπάρχουν τέλη στην περίπτωση της ελικτότητας και η Σάρον νομίζω και ο Μπούρχαρ έχουν υποβάλει σχετικές τροπολογίες και επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις ε, να ε, επιτρέπεται η προσωρινή αναστολή μονάδων ε, και μετοχών. Προσέξαμε ότι και άλλοι έχουν υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Η όλη συζήτηση σχετικά με τη διατήρηση των ΣΥΝΑΒ και τις εναλλακτικές προτάσεις δεν αποτελεί απάντηση ε, στο πλεονέκτημα του first mover. Και δεν έχω βρει κάποια σωστή αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Επίσης, ε, προϋποθέσεις μεταβατικής περίοδου. Και εμείς στηρίζουμε απολύτως ε, τον εισηγητή στην ε, απαγόρευση των φορολογικών ε, παραδείσων. Ε, αναγνωρίζω εδώ κάποια διατύπωση που έχω δει αλλού. Επίσης θέλουμε να προστατεύσουμε το χρήμα του φορολογούμενου πολίτη. Επίσης απαγορεύουμε την εξωτερική υποστήριξη από διάφορες περιφερειακές τοπικές αρχές κλπ. Επίσης, όσον αφορά τα παράγωγα, Θέλουμε να περιοριστεί η επένδυση ε, σε παράγωγα τα οποία να εμπορεύονται σε ρυθμισμένη αγορά. Αναγνωρίζω και την πτυχή των MIFID και ο Ζαμπόλ προτείνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή και προτείνουμε επίσης ε, να ρυθμιστεί η πολιτική αμοιβή. του ε, MMF και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε διαφορετικές πολιτικές ε, αμοιβή. Ελπίζω το δικαστήριο πάντως να συνεχίσει να, να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση και να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να νομοθετεί στους τομείς αυτούς. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την ε, ΕΑΚΑ το οποίο σημαίνει ότι τα ε, συστημικά αμοιβαία κεφάλαια του, της χρηματογοράς να ελέγχονται από την ε, ΕΑΚΑ. Επίσης προτείνουμε τα αμοιβαία κεφάλαια της ε, χρηματαγοράς να αναγκάζονται να έχουν προγράμματα αποκατάστασης σε περίπτωση που βρίσκονται υπό πίεση. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο, ακόμα και αν ε, είναι επιτυχές μόνο κατά 80% είναι καλύτερο από το να μην υπάρχει τίποτα. Θα κλείσω εδώ και προσβλέπω στην ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση, και, η οποία νομίζω ότι θα είναι και έντονη, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε εξετάσει μόνο τα εύκολα κομμάτια του κειμένου. Φαντάζομαι ότι θα προχωρήσουμε σύντομα στα πιο δύσκολα μέρη. Προσβλέπω στην καλή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρέτσακ και πάλι έγινε Σαΐτ Καλημέρα σας και πάλι. Εξ ονόματος του Σατζίτ Καμάλ. Ε, <clears throat> ναι, έχει μερικά σχόλια να κάνει. Θέλει να ευχαριστήσει τον Σίγητη ε, και τους Κιώδη για την καλή συζήτηση όσο και παραγωγική που είχαν χτες. Ωστόσο, θα ήθελε και πάλι να τονίσει και να επαναλάβει τη θέση του ε, για το αποθεματικό των σταθερών καθαρών αξιών ενεργητικού ΣΥΝΑΦ. Το 2008 ε, η μαζική ε, κατάσταση που δείξει σε αυτό είχε να κάνει με την υπερβολική έκθεση στον Αμερικανικό τομέα. Το αναγνώρισε αυτό το 2012 σε μια έκθεση της ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροφή, ότι οι σταθερές και οι κειμενόμενες και η ΣΥΝΑΦ και η ΒΙΝΑΦ αμοιβαίων κεφαλαίων δεν ήταν οι ε, σωστές ε, αξίες. Οι κεφαλαιακές ε, απαιτήσει έχουν σχεδιαστεί για τράπεζες, όχι για τέτοια κεφάλαια και δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα ώστε να είναι βιώσιμα αυτά τα κεφάλαια. Ε, διάφορες τοπικές αρχές, ε, φιλανθρωπικά ιδρύματα, σωματεία, κάθε είδους ε, ενδιαφερομένοι απευθύνθηκαν στον κύριο Καμάλ και οι ίδιοι διαχειριστές τέτοιων ταμείων και θεωρούν ότι το αποθεματικό ασφαλείας είναι μέγα σφάλμα. Το buffer μπορεί να το ζητούν οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, αλλά υπάρχει διαφωνία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των εποπτών ε, κινητών αξιών. Δεν χρειάζεται 3% αποθεματικό. Θα πρέπει να ε, υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τα τέλη και τις προσβάσεις. Αν θέλουμε ε, να έχουμε καλύτερες λειτουργίες, καλύτερη λειτουργία της αγοράς αξιών, πρέπει να σχεδιάσουμε διαφορετικά το αποθεματικό ασφαλεία σε διαφορετικό ε, πλαίσιο. Ε, το buffer, το αποθεματικό ασφαλείας θα σκοτώσει ε, τις κειμενόμενες αξίες, τα βίνα. Αν αυτό θέλετε, να το πείτε όμως και να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους επενδυτές διαφόρων κατηγοριών για να κανονίσουν την πορεία τους και να προετοιμαστούν για αυτή την κατάσταση. Αυτά είπε ο κύριος Καμάλ, διαστόματος του κυρίου Στρέιτσεκ ο Γκέι Μίτσελ, η Σιλβί Γκουλάρ, επόμενη Αστρίτ Λούλινγκ και η Ομιλούσα. Άλλου παρόντε βουλευτέ δεν είναι. Α, έχουμε. Α, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει κανεί το λόγο, θα το ξαναπούμε αργότερα. Γκέι Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του Σκιώδη. Ο Ζαν Πολ έχει δίκιο. Υπάρχουν διεστάμενε απόψει, ιδιαίτερα όσον αφορά τι σταθερέ ΚΑΕ. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό. χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Γενικά στηρίζω την ε, προσέγγιση αυτή. Μου έκανε εντύπωση κατά την ε, επίσκεψη στην Ιρλανδία τις προηγούμενες εβδομάδες ε, που ένας Ιρλανδός βουλευτής αναφέρθηκε στους κατόχους ομολόγων ότι θα έπρεπε να είχαμε κάψει τα ομόλογα και να δούμε τι θα γινότανε. Νομίζω ότι κινδυνεύουμε εάν ε, καταργήσουμε την δυνατότητα να υπάρχουν σταθερές ε, ΚΑΕ. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να εξαλείψουμε τους κινδύνους ε, για τους συστημικούς κινδύνους, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Οι συμβουλές που μου έδωσαν εμένα είναι ότι ιδιαίτερα το αποθεματικό ασφαλείας θα στρεβλώσει την ρευστότητα με μη προβλέψιμους τρόπους. Και θα δούμε ε, φυγή προς την ρευστότητα κεφαλαίων και αυτό δεν ε, θα το θέλαμε. Στην Ιρλανδία έχουμε πρόβλημα με τις καταθέσεις. Είναι δύσκολο το, να κάνουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί με επικοδομητικό τρόπο τα κεφάλαια. Μπορούμε λοιπόν να δούμε να μεταφέρεται η ρευστότητα εκτό τη Ευρωπαϊκής Ένωση και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι σταθερές ΚΑΕ αποτελούν τεράστιο μέρος ε, της ε, ρευστότητα του επιχειρηματικού τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τις ε, ρυθμιστικές διαφορές ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Επίσης ε, άκουσα για το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Στο σημείο 12.1 ε, μας έδωσαν διαφορετική εντύπωση για τις ε, σταθερές ΚΑΕ από αυτή που ακούμε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να πω ότι είπε ο Επίτροπος Κάλαχερ που είπε ότι, δεν, ότι οι δικοί μας οικονομολόγοι πιστεύουν ότι ένα αποθεματικό ασφαλείας ε, για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλο και δεν θα επιτρέψει στα μηδέα κεφάλαια να λειτουργούν. Εάν είναι τόσο μικρό ώστε να ε, αξίζει οικονομικά τον κόπο δεν θα αποτελεί καμία προστασία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θα ήθελα να πω το εξή. Δεν θέλει μόνο ο χρηματοοικονομικός τομέας ε, να περάσει εύκολα. Αυτό είναι σημαντικό θέμα για τον οικονομικό τομέα γενικά, για τη βιομηχανία. Ακούστε τι λένε οι επενδυτές, ε, τι λένε οι οικονομολόγοι. Είχαμε πρόσφατα μία συνάντηση με πανεπιστήμια, με στεγαστικούς οργανισμούς, με τοπικές αρχές ε, που λένε ότι θέλουμε ε, ρευστότητα, φερεγγιότητα και απόδοση. Φερεγγιότητα, ρευστότητα, απόδοση με αυτή τη σειρά. Και εάν καταργηθεί αυτό δεν θα έχουμε καμία εναλλακτική λύση και θα πρέπει να το σκεφτούμε. Όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους, που νομίζω ότι είναι αρκετά απόμακροι, νομίζω ότι τα τέλη ρευστότητα ε, θα αποτελέσουν έναν συμβιβασμό με τον οποίο μπορούμε να καλύψουμε τις ε, σχετικές ανησυχίες. Πρόεδρε, δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά μας ανησυχεί το θέμα αυτό. Νομίζουμε ότι είναι επικίνδυνο πεδίο και δεν θα ήταν σοφό να μην συνεχίσουμε να έχουμε και, τα, και τις σταθερές ΚΑΕ και τις κειμενόμενες. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να βλάψει την Ευρώπη. Και έτσι να δώσουμε μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις ΗΠΑ και άλλους. Ας συνεργαστούμε λοιπόν για να έχουμε ένα λογικό αποτέλεσμα, όπως κάνουμε πάντα. Θα ήθελα να καλέσω τους ευρωβουλευτές ε, να μην κάψουμε τα, χλωρά μαζί με τα, ξε... τα ξερά μαζί με τα χλωρά, τα χλωρά μαζί με τα ξερά, ε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για την ρευστότητα και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους εσκιώτης για τη δουλειά που έχουν κάνει πάνω στο δύσκολο αυτό θέμα. Ευχαριστώ, Σιλβί. Ευχαριστώ, Σάρων. Συμφωνώ, μάλλον συμμερίζομαι ε, τον προβληματισμό του Κάι, γιατί πραγματικά... Ε, αντιπροσωπεύουν πολλά εκατομμύρια που είναι απαραίτητα για την ρευστότητα της αγοράς. Εγώ δεν λέω ότι ε, θα πρέπει στην Ευρώπη να περάσουμε από την τραπεζική χρηματοδότηση στη χρηματοδότηση μέσα από τις αγορές. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα σημείο επί του οποίου υπάρχουν ε, πολλές διαφορετικές απόψεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων και εγώ χωρίς να λέω ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια, λέω, λέω ότι υπάρχουν ε, κάποια εργαλεία τα οποία μαζικά χρηματοδοτούν την Ευρωζώνη και που επομένως ίσως θα έπρεπε να δούμε το ενδεχόμενο να τα ε, χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από ό,τι άλλο να είναι προτιμότερα ας πούμε. Ε, όσον αφορά τώρα τα σταθερακά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια, ε, κάποια στοιχεία προστασίας, κάποια buffers δεν ξέρω αν σας πολύ βοηθάει αυτό που σας λέω κύριε εισηγητά Ωστόσο να ξέρετε ότι είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι να δούμε από πολύ κοντά να μελετήσουμε τις συμβαστικές σας προτάσεις. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε τις συγκρίσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί έχουμε άλλη δομή αγορών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Astrid. Merci, madame. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά την παρέμβαση του συναδέλφου Μίτσελ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Συμφωνώ πολύ με τα όσα είπε προσωπικά κατά την ε, πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα που είναι σημαντικό εργαλείο επενδύσεων και για τους θεσμικούς επενδυτές αλλά και για τους μικροεπενδυτές. Κάναμε αυτή τη συζήτηση λοιπόν και είχα κάνει ευθύ εξ αρχής δύο σχόλια και πιστεύω ότι αυτά τα σχόλια διατηρούν ε, την εγκυρότητα τους ε, στο ακέραιο βρισκόμαστε σήμερα σε ένα περιβάλλον που καθιστά τα πράγματα πάρα πολύ ευαίσθητα με επιτόκια που σχεδόν φτάνουν στο μηδέν. Είναι πάρα πολύ λεπτή η κατάσταση για πάρα πολλούς φορείς. Ε τις χρηματαγοράς, οι αποδόσεις και τα περιθώρια που έχουν ε, οι ε, επαγγελματίες είναι τόσο συμπιεσμένα που οποιαδήποτε αλλαγή του κανονισμού ή της νομοθεσίας θα έχει τεράστιες επιπτώσεις. Εάν τα επιτόκια ε, της τάξης του 5-6% ήταν 5-6% θα ήταν ε, αμεληταία μια διαφορά της τάξης του ε, ενός τετάρτου της ποσοστίας μονάδας. Αλλά όταν είναι μισό της και η 0,25 τα επιτόκια καταλαβαίνουμε ότι είναι ζωτική σημασία και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για το τι αποφασίζουμε. Ένα δεύτερο είναι ένα πάγιο επιχείρημα. Ε, για την λογιστική καταγραφή του κόστους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να αλλάξει βάθρων τους κανόνες. Προτείνει ένα είδος αποθεματικό ασφαλείας στο buffer 3% απαντάει ο κλάδος λέγοντας ότι Μα τι είναι αυτό, έκτακτος φόρος. Αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να το δούμε. Εγώ θα ε, ήθελα να πω ότι τα συνάβη σταθερές καθαρές αξίες ενεργητικού θα πρέπει να είναι μόνο για θεσμικούς επενδυτές. Μου λέγουν ότι δεν έχει ρυθμιστεί επαρκώς αυτό ακόμα. Μα γιατί να μην διαλέξουμε αυτή την κατεύθυνση. Όταν έχουμε θεσμικούς επενδυτές, αυτοί δεν πρόκειται να ε, κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις τύπου RUN και ε, ασυντόνιστες και Επίσης, σε ό,τι αφορά και πάλι το πλαίσιο των πολύ χαμηλών επιτοκίων, εγώ θα ήθελα να σβήσουμε το Μπάφερ ε, το αποθεματικό ασφαλεία Δεν είναι θέμα του νομοθέτη τώρα να δυσκολεύει τη βιωσιμότητα ενός χρηματοοικονομικού μέσου που έχει αποδειχθεί χρήσιμο και ωφέλιμο στην πράξη και απομένει να αποδειχθεί η επικινδυνότητά του και το ρίσκο του. Εγώ πιστεύω ότι οι ε, αποδείξεις που μας δίνεται δεν είναι αρκετά πιστικές για να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Εμείς ε, όλο ζητούμε και διεκδικούμε περισσότερη απασχόληση, περισσότερη ανάπτυξη της οικονομίας. Ε, τώρα γιατί θέλουμε να ρυθμίσουμε κάτι που θα διώξει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις οποίες χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Ελπίζω και στη δική μου πολιτική ομάδα να πριτανεύσει η λογική τελικά. Thank you uh, Ευχαριστώ πολύ. Μπέρκαρτ έχει ζητήσει το λόγο. Κύριος Μπάλτς, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πολύ σύντομα ε, θα ήθελα να παρουσιάσω μερικά στοιχεία από πλευράς μου. Παρόλο που σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, ε, Γκέι Μίτσελ και με την Άστριτ Λούλινγκ. Στο θέμα αυτό του αποθεματικού ασφαλείας, το buffer, είμαι ε, σαφέστατα υπέρ της διαγραφής αυτού, διότι αν κάνουμε ένα τέτοιο buffer αποθεματικού ασφαλείας, τότε ε, θα διακυβεύαμε το σύνολο των σύναυς των σταθερών καθαρών αξιών ενεργητικού. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργούσε καν μια τέτοια αγορά, διότι δεν θα ήταν σκόπιμη από πλευρά κερδοφορία. Τώρα, κατά πόσο οι σταθερέ θα γίνουν κειμενόμενε, τα σύναυσα, βίναυς. Ε, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Εντάξει, να γίνει μια ε, τροποποίηση, μια, μια μετάβαση, αλλά όχι αυτόματα. Θα πρέπει να είναι δεδομένη η εποπτεία, όπου χρειάζεται αυτό πάντα και όπου είναι και εφικτό και αποδεικνύεται στην πράξη λειτουργικό. Ακούσαμε και για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Αμερικανικές Εποπτικές Αρχές ε, μόλις έκαναν μια διαβούλευση για τη ρύθμιση των ε, αξιών αυτών περιμένουν να γίνει αυτό σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών τους επόμενους μήνες. Εμείς δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε τους Αμερικανούς, έχουμε και δικές μας ανάγκες. Να καθίσουμε να σκεφτούμε κατά πόσο μας εξυπηρετεί ο ρυθμός που έχουμε επιλέξει, γιατί έχουμε και εμείς ε, υποχρεώσεις απέναντι στο G20. Και ένα τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι οι κανόνες για τις καταθέσεις και για τη διαφοροποίηση των προϊόντων. Ε, δεν χρειάζεται να ε, κρυβόμαστε. Ε, η κρίση μας έδειξε ότι υπήρξαν ε, ανεπάρκειες, γι' αυτό χρειάζεται ρύθμιση χωρίς υπεκφυγές να το λέμε και να ελέγχουμε στο μέλλον και να εξασφαλίζουμε την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των αξιών. Εγώ έχω κάποιες επικρίσεις για διάφορα πράγματα, γι' αυτό και πρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα των διαφόρων προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Είπα και εγώ ότι ήθελα να εγγραφώ για να μιλήσω, αλλά θα πω δυο λόγια και μετά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόνα. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι όσον αφορά τις σταθερές ΚΑΕ, σύναψη. Ε, ξέρουμε ότι ε, το θέμα είναι να ε, βρούμε λύση όσον αφορά και τα αποθεματικά ασφαλείας και όσον αφορά τη διαφάνεια. Ε, βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε και την εξωτερική αξιολόγηση ε, μαζί με τις εσωτερικές διαδικασίες ε, αξιολόγησης. Και εδώ οι απαιτήσει ασφαλεία και διαφάνειας θα πρέπει να είναι ε, πιο απαιτητικές. Όσον αφορά τα σύναυσα και ο Μάριο Ντράγκη και η Ένωση Κεντρικών Τραπεζών έχουν ε, ε, κάνει σχόλια σχετικά. Από όσο καταλαβαίνω βασίζονται ε, στην αρχική αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν. Όμως το αρχικό δείγμα ε, της, ε, δι, της μελέτης ε, τελικά ήταν περισσότερο σε βίναυς, σε κειμενόμενες αξίες και επομένως τα αποτελέσματα ενδεχομένως αυτό το 1% όσον αφορά τους θεσμικούς επενδυτές να μην είναι πολύ σωστά και όπως υπόθηκε προηγουμένως και για τις συνεταιριστικές διατηρητικές επενδυτικές αρχές αλλά και για άλλους είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις ε, ροές που ξεπερνούν το 1% ε, σε διάρκεια τριών ε, ημερών αλλά σε γενικές γραμμές αυτά ειδικά στο short selling γίνονται συνέχεια και χρησιμοποιούνται πάρα πολύ από τις συνεταιριστικές αρχές έτσι ώστε να λύσουν τα καθημερινά προβλήματα ρευστότητας. Αυτό που λένε δηλαδή business as usual, αλλά θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει ακριβώς. Επίσης, ε, όσον αφορά τις μικρές ε, ε, εταιρείες ε, φιλανθρωπικές και τα λοιπά. Ε, αυτά ίσως μπαίνουν στο μύφιντα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να, μην, να μην αποτρέψουμε παντελώς τους μικρούς επενδυτές να χρησιμοποιούν αυτά τα ε, εργαλεία. Από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε καθαροί. είτε, δηλαδή, τα χρήματα τα οποία δεν μπαίνουν σε αυτές τις επενδύσεις δεν μπαίνουν, και δεν μπαίνουν στα ΣΥΝΑΒ δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι πηγαίνουν ε, στα, στα ΒΙΝΑΒ, στις ε, ε, κειμενόμενες ε, καθαρές αξίες ενεργητικού. Θα πρέπει να τα δούμε. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ε, ε, κάνει και το πρόγραμμα προστασίας καταθέσεων. Η Ιρλανδία έπρεπε να, να εγγυηθεί όλες τις καταθέσεις ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ζημιογόνο. Απ' την άλλη πλευρά ε, ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποια όρια όσον αφορά την εγγύηση των καταθέσεων στις τραπέζεις και εάν δούμε, βλέποντας από κοντά την ιεραρχία αυτών των διασώσεων που έχουν γίνει, των bailout, πραγματικά ε, είναι αναγκαίο να μην πάνε τα χρήματα αυτά στις τράπεζες. ενδεχομένως ε, τα funds αυτά δεν λειτουργήσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά η λύση ε, δεν είναι να τα καταργήσουμε, ε, είναι να παραδεχτούμε ότι ορισμένα πράγματα δεν λειτουργήσαν όπως τα θέλαμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα του παρελθόντος έτσι ώστε να γίνουν πιο σωστές όλες οι κινήσεις μας. Ε, όσον αφορά τώρα τα, τη διασφάλιση της ρευστότητα μίας ημέρας και 15 ημερών, ειδικά για τους εθνικούς επενδυτές, θα πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, θα αναφερθώ στις τάσεις ε, φυγής, τα runs και θα αναφερθώ και στα τέλη ρευστότητα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι η τάση για φυγή μπορεί να υπάρχει και στις σταθερές και στις κειμενόμενες ε, ΚΑΕ σε περίπτωση κάποιου πιστοτικού συμβάντος ή κάποια πιθανή κρίση σε κάποιον τομέα, ιδιαίτερα τον τραπεζικό. Υπάρχει όμως ε, μια σημαντική διαφορά. Σε περίπτωση σταθερής ε, ΚΑΕ υπάρχει ένα θέμα σταθερότητας ε, που δεν έχουν κειμενόμενες. Ε, δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε τον πυρήνα της πρότασης μας που είναι η ρευστότητα. Επίσης η δεύτερη αρχή είναι το μοίρασμα των κινδύνων. Σε περίπτωση φυγή είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά... Οι σταθερές έχουν ένα επιπλέον πρόβλημα σταθερότητας. Θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποιο αποθεματικό ασφαλείας ε, για να τη στήριξει. Είπαμε ότι μπορεί να αντικατασταθεί το μπάφερα από ε, τέλη ρευστότητας, κάτι που λειτουργεί σαν αποθεματικό ασφαλείας επειδή πληρώνει κανείς κάποιο επιπλέον ποσό. Και αυτό είναι αλήθεια εάν είναι μόνιμο μέτρο. Ε, αυτό το τέλος. Εάν είναι προσωρινό αυτό δεν ε, ισχύει και η κρίση έδειξε ότι τη στιγμή ε, που υπάρχει η δυνατότητα του sponsorship κανένα κεφάλαιο δεν θα δεν θα απελευθερώσει τα τέλη ρευστότητα, διότι δεν θα θέλουν να ομολογήσουν ότι κοντεύουν να πέσουν κάτω από την τιμή αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Right, that's the end of the speakers. Um, Ευχαριστώ. Ο εισηγητής θέλει το λόγο ε, για να συνοψίσει. Ναι, πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα όσα είπανε. Και εγώ είχα πει ότι είναι πολλά τα σημεία που συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Υπάρχουν κάποια κρίσιμα ε, τι θα κάνουμε με τα σύναυση σταθερές καθαρές αξίες ενεργητικού. Χρειάζεται συζήτηση εκεί. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να βρούμε κάποια συνένεση. Θα κάνω ό,τι μπορώ τουλάχιστον ό,τι περνάει από το χέρι μου εμένα. Θα ήθελα να διορθώσω κάτι. Ότι οι συστάσεις είναι παλιές. Ε, μα το 2013 είναι. Δεν είναι και τόσο παλιές. Ο κύριος Ντράγκη ήρθε εδώ τον Οκτώβριο και μας είπε ότι είναι υπέρμαχος του να φύγουμε από τις αφαιρές αξίες και να πάμε στι Όχι σύννεφα αλλά βίναφ. Σε ό,τι αφορά τον buffer, το αποθεματικό ασφαλείας, υπάρχουν πολλές μελέτες που το ζητούν. Διάβασα τη μελέτη που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, όπως σας είπα το Δεκέμβριο του 2013. Θα τη στείλω και στους κοιόδες ε, για να μπορέσουν να εξοικειωθούν. Αυτά. Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε με τους κοιόδησιητές ε, για να ε, συντονιστούμε ακόμα περισσότερο και ελπίζω το Φεβρουάριο να έρθει και η ψηφοφορία έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα. Για εκείνους που λέγουν ότι α, περίμενε να αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τι θα κάνουν και, και εκείνοι. Θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς να περιμένουμε εκείνοι εμάς να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Για ποιο λόγο να περιμένουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας καθοδηγήσουν. Εμείς να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε για να κάνουμε μια καλή νομοθεσία και από εκεί και πέρα προσπαθώ εγώ πάντα και συνεχώς ως εισηγητής να έχω επαφές και με τους συναδελφούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, να παρακολουθώ τις εξελίξεις, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει εμείς αναγκαστικά να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. So, uh... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν μπορούμε θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε στις 12 Φεβρουαρίου ακόμα για να πάει στην Ολομέλεια του Απριλίου. Τον Απρίλιο όλη μέρα θα ψηφίζουμε, κάθε μέρα. Με αυτό το ρυθμό που πάμε, ε, προετοιμαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στο σημείο που είναι το επόμενο και δεν είναι το 12 γιατί έχει να βληθεί. Θα πάμε στο σημείο 13, Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια και πάλι οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, η συγγήτρια και η σκιώδης είναι παρόντες, εξέταση των τροπολογιών της έκθεσης κυρίας Ρόδη Κράτσα. Θα δώσω το λόγο στη Ρόδη. Παρακαλώ κύριε Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους για την, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους σε αυτό το, αυτή την έκθεση. Ε, κατατέθηκαν 294 τροπολογίες, μεταξύ αυτών είναι και κάποιες δικές μου. Και όπως ξέρετε προβλέπεται η τελική ψηφοφορία στις 17 Φεβρουαρίου. Θα κάνω μια πρώτη ε, προσέγγιση σήμερα των τροπολογιών και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα έχουμε επί της ουσίας ε, και συγκεκριμένων προτάσεων μια συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Καταρχάς ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τους συναδέλφους είναι εάν στο ταμείο αυτό ε, μπορούν να ε, συμπεριληφθούν οι εισηγμένες εταιρείες ε, ποιες εταιρείες μπορούν να περιληφθούν στο 70% των επιλέξιμων κεφαλαίων. Ε, κάποιες τροπολογίες περιορίζονται στις εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες εννοώ με βάση τον ορισμό της Επιτροπής. Άλλες τροπολογίες ε, στοχεύουν σε εισηγμένες με κεφαλοποίηση έως ένα δισεκατομμύρια ευρώ ε, που είναι μεγαλύτερο το επίπεδο από αυτό του ορισμού της Επιτροπής και άλλες είναι να, τροπολογίες αναφέρονται στο να όλες οι εισηγμένες εταιρείε να αποτελούν επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία. Ε, το ζήτημα τώρα είναι ποιες ε, από αυτές τις εισηγμένες επιχειρήσεις ε, μπορούμε να επιλέξουμε, διότι γενικά είναι έντονο το αίτημα της συμπερίληψης των εισηγμένων, αλλά ποιες, ποιες επιχειρήσεις από τις εισηγμένες. Η δική μου άποψη είναι να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εισηγμένες, διότι είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από ρευστότητα και έχουν ανάγκη να βρουν ε, πόρους. Θα ακούσουμε συνέχεια και την άποψη των εισηγητών. Άλλο κρίσιμο θέμα ε, των, εννοώ, όχι των, των σκιωδών εισηγητών και των συναδέλφων. Άλλο κρίσιμο θέμα είναι ε, τα δικαιώματα εξαγοράς. Μέσα στην προσπάθεια ε, του να γίνει ελκυστικό το νέο αυτό εργαλείο υπάρχει η, αντίληψη ε, της δυνατότητας, να δοθεί δυνατότητα εξαγοράς ε, δικαιωμάτων διότι υπάρχει πάντα η δυσκολία του να αισθάνονται δεσμευμένοι οι άνθρωποι μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του Ταμείου. Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις, ε, τρεις μάλλον. Από τη μια μεριά είναι ε, να μην δοθεί κανένα δικαίωμα εξαγοράς για να υποστηριχθεί ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της προσπάθειας. Απ' την άλλη είναι να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς σε όλους τους επενδυτές, θεσμικούς, μη θεσμικούς, για να, ιδιώτες, για να είναι πιο ελκυστικό το εργαλείο αυτό. Και από την άλλη πλευρά είναι μια μέση οδός ε, το να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς μόνο σε ιδιώτες επενδυτές και μάλιστα υπό προϋποθέσεις. Εκεί καταλήγει και ε, η δική μου πρόταση. Ε, μια ενδιαφέρουσα πρόταση έχει κάνει και ο Ζαν Πολ για τις δυνατότητες μείωσης του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ΕΜΕΚ, που καταλα... του, του ταμείου αυτού, που καταλαβαίνω ότι εννοεί ε, τη δυνατότητα του να μπορεί να βγει κάποιος από το περιουσιακά στοιχεία. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας το εξηγήσει μετά ο Ζαν Πολ. Ε, άλλο θέμα κεντρικό είναι ο κύκλος ζωής. Ε, έχω προβληματιστεί και εγώ και συνάδελφοι πώς μπορεί να οριστεί αυτός ο κύκλος ζωής χρονικά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να, δεν έχει νόημα να συνεχίσει όσο, όπως έχει προβλεφθεί το Ταμείο και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου κάνει μια ενδιαφέρουσα επένδυση με προοπτικές και αξίζει να παραταθεί ο κύκλος ζωής. Ε, είναι λοιπόν ένα κρίσιμο ερώτημα πώς θα κρατήσουμε το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα όπου πρέπει να έχει ένα κύκλο ζωής, δεν μπορεί να είναι για λίγα, πολύ λίγα χρόνια, πώς θα είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τι προοπτικές δίνουν τα περιουσιακά στοιχεία και πώς ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα με τη σύμφωνη γνώμη των επενδυτών, σημειώνουν ε, με του συνάδελφοι, θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την λήξη ή την παράταση του κύκλου ζωής. Ε, άλλο, άλλο θέμα που απασχολεί μέσω τροπολογιών, το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε, δεν έχω καταλήξει κι εγώ απόλυτα, είναι στο να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν επαγγελματικά ταμεία, τα οποία θα έλξουν ευκολότερα τους θεσμικούς επενδυτές ε, και ε, ε, που θα απευθύνονται σε μικρότερο βαθμό σε ιδιώτες επενδυτές. Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι δεν μπορούν να συνεπάρξουν μαζί οι επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές διότι έχουν διαφορετικές γνώσεις, διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετικούς στόχους. Ότι είναι δύο ομάδες που θα πρέπει να έχουν καθένα το ταμείο του. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το συζητήσω με τους συναδέλφους. Ε, μια, ένα άλλο θέμα που έχουμε θέσει είναι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση των επενδύσεων ε, εγώ προτείνω να έχουμε ένα συνδυασμό ε, οπωσδήποτε βάσης 60-40, δηλαδή το 60% να επενδύονται σε έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 40% να είναι έξω. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση του να είναι 50-50. Δεν το θεωρώ ο, ε, ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο διότι όλα εξαρτώνται από την αγορά, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή και την επίτευξη ε, αφενός των στόχων της ενίσχυσης των υποδομών και της αγοράς στην Ευρώπη αφετέρου και του κέρδους. Οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε αν και προτείνω ε, κατά λίγο να κρατήσουμε το 60-40. Ε, άλλες τροπολογίες έχουμε τις μεγαλύτερες δυνατότητες δανεισμού για τα ταμεία αυτά ε, έως 40% αντί του 30% που προτείνει η Επιτροπή. Και δεν είμαι ε, πολύ υπέρ αυτής της, ε, της πρότασης. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να κρατήσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Ε, έχουμε άλλες τροπολογίες για, την ενίσχυση των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίωσης του κανονισμού ε, δεν ξέρω το άπαξ και ήδη προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες μου φαίνονται ότι είναι ε, ικανοποιητικές. Ε, μετά στα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία έχουμε κάποιες ε, επίσης τροπολογίες. Ε, άλλοι συνάδελφοι σκέπτονται να α, μη συμπεριλαμβάνεται το real estate, τα περιουσιακά στοιχεία από το real estate ενώ άλλοι συνάδελφοι ζητούν να συμπεριληφθούν και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε ε, να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Ε, άλλο ο θέμα είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντολογικών και των κοινωνικών κριτηρίων. Πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να γίνουμε περισσότερο δεσμευτικοί στον τομέα αυτό διότι τα περιβαλλοντολογικά κριτήρια έχουμε μια ισχυρή νομοθεσία την οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Ως προς τα κοινωνικά κριτήρια ε, και αυτά εμπεριέχονται αλλά δεν είναι και το αντικείμενο και ο κεντρικός, βασικός στόχος του, του ταμείου αυτού του οποίου ε, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές ε, η, η αποτύπωση των τροπολογιών και των και των ε, αν θέλετε, απόψεων που έχουν εκφραστεί και περιμένω την άποψη των συναδέλφων προτού καταλήξουμε στην, ε, στους συμβιβασμούς και στις προτάσεις για την ε, συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Right. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ ο Σαΐντα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισαγωγή της και για το έργο της γενικότερα. Βεβαίως περιμένουμε περισσότερο το σχέδιο των συμβιβασμών και αυτή τη στιγμή θα το έχουμε ε, το κείμενο, θα μπορέσουμε να κάνουμε συζητήσεις και να προχωρήσουμε. Γενικά υποστηρίζουμε βεβαίως την πρόταση μακροπρόθεσμα ε, επενδυτικά κεφάλαια να δημιουργηθούν. Θα πρέπει να βρούμε όμως έναν τρόπο και δεν είμαι ο μοναδικός που το λέω. Ε, ε, ούτε ο μοναδικός τόπος να ενισχύσουμε την οικονομία αλλά να ξεφύγουμε λίγο από την εξάρτηση από την τραπεζική χρηματοδότηση. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ουσιαστικά έργα υποδομών και γνήσια δεν είμαστε υπέρ το να ε, το συνδέσουμε αυτό με το real estate, ε, με τα ακίνητα. Υπάρχουν άλλα εργαλεία γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση, συμφωνούμε ότι μπορεί να είναι ε, μια σημαντική τεχνική, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι με τρόπο διαφανή και καλά πλαισιωμένη η διαμόρφωση. Η συζήτηση για τον κύκλο ζωής τώρα του Ταμείου το κεφαλαίο αυτό είναι κάτι που συνδέεται με τον επενδυτή. Αν είναι θεσμικός ή αν είναι μικροεπενδυτής ηλιανικής, ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, θεσπίσουμε σαφείς κανόνες για το πώς μπορεί κανείς να βγαίνει από ένα τέτοιο κεφάλαιο, αλλά δεν θα πρέπει να ε, διακινδυνευθεί η εξασφάλιση των μέλλον των επενδύσεων ή του έργου για το οποίο έχει μπει κανεί σε αυτό το κεφάλαιο όταν θέλει να φύγει. Γι' αυτό μιλούμε για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Και όταν κάποιος μπαίνει σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει και συνέπειες, ότι είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Υπάρχουν διάφορα σημεία που θα πρέπει να λύσουμε και για μας είναι κρίσιμα αυτό που σας ανέφερα. Ε, Ευχαριστώ. Α, εσύ θα πάρει τον λόγο. Ναι, ναι. Θα μιλήσω εξ ονόματος του Ντεμπάκερ, ο οποίος ζητεί συγγνώμη γιατί κολλείεται. Θα διαβάσω αυτά που μου ε, ε, έδωσε. Δεν μπόρεσα να συζητήσω προσωπικά μαζί του. Θα διαβάσω λοιπόν. Ήδη στι άλλες δύο συζητήσεις ε, για το θέμα αυτό ε, είπε ότι καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και γενικές γραμμές είναι υπέρ. Ε, υπάρχει ένα equity gap το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί έτσι ώστε να, η ανάπτυξη η οποία θα προωθηθεί να είναι βιώσιμη από κάθε άποψη. Επίσης είναι ο βαθμός εξάρτησης από την τραπεζική χρηματοδότηση πολύ μεγάλος και επομένως θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση. Ωστόσο, ο κύριος Ντεμπάκερ λέει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι υπάρχει έλλειψη μακροπρόθεσμης ε, χρηματοδότησης, ε, ενώ ε, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Η έλλειψη της μακροχρόνιας χρηματοδότησης ερώτησης. Ίσως σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να λυθεί μέσω της αγοράς, αλλά ε, υπάρχουν ε, ε, πολλές νομοθεσίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Παράδειγμα, στην συζήτηση για τα ΠΡΙΚΠ συζητήθηκε το θέμα της περίπλοκης νομοθεσίας και πρέπει να βρεθούν λύσεις απλούστευσης της νομοθεσίας που δεν θα ισχύει όμως για την λιανική ε, τραπεζική χρηματοδότηση. Επίσης, όπως προτείνεται η νομοθεσία, χρησιμοποιεί ένα μέτρο για όλους, one size fits all, ενώ υπάρχουν μεγάλες, μεγάλοι επενδυτές μικρότεροι, υπάρχουν μεγάλες εταιρείε, μικρότερες, μεσές κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν διαφοροποιημένη ε, προσέγγιση έτσι ώστε να καλύπτονται καλύτερα τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα όλων. Ε, θα υπάρξουν τροπολογίες από την πλευρά ε, Debaker. Ε, έτσι ώστε να ε, είναι πιο ε, καθαρά ορισμένες οι κατηγορίες, αν θα είναι ανοιχτέ για όλους, αν θα είναι μόνο για ορισμένους επενδυτές, επαγγελματίες επενδυτές, αν θα είναι open-ended κτλ. Ελπίζουμε ότι η συγγήτρια θα λάβει υπόψη τις τροπολογίες μας και φυσικά πάντοτε θα είμαστε στη διάθεση όλων για ε, συζήτηση. Αυτά μου έγραψε ο κύριος ε, Ντεμπέκερ και θα το δώσω και στην συγγήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Φιλίπ, ε, εσύ ξανά για τους πράσινους. Ναι, είναι η μέρα που παίζω πολύ. Μας αρέσει η πρόταση της Επιτροπής ως έχει, ε, διότι στην ουσία ε, δίνει στους ε, υπομονητικούς επενδυτές τρόπους επένδυσης. Επομένως, επομένως αυτές οι ανησυχίες για αλλαγή του στόχου της νομοθεσίας αυτής δεν μας βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Εδώ υπάρχει επιβράβευση των υπομονετικών. Ε, συμφωνούμε λοιπόν γενικά με την Κομισιόν. Θέλουμε απλώς να διασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσει ε, οι οποίες εισάγονται δια της νομοθεσίας αυτής ε, είναι αρκετά λογική και αρκετά φιλόδοξη, αλλά ωστόσο να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Έχουμε κάποιες τροπολογίες, δεν θα ασχοληθώ με όλες, αλλά με ορισμένες από αυτές. Θέλουμε βεβαίως η πληροφόρηση να είναι ε, πιο καλή και από την αρχή 136, 146, 137 και επίσης θέλουμε πληροφόρηση για την εξέλιξη ε, της επένδυσης και του κόστους. Επίσης θέλουμε ε, η ποιότητα να είναι σωστή, γιατί εδώ αναφερόμαστε και στους διαχειριστές. Ε, θέλουμε ε, να υπάρχουν κάποιες νομικές δεσμεύσεις, να μην έχει υπάρξει για αυτούς απαγόρευση διανόμου κτλ. κτλ. Να έχουν δηλαδή τα απαραίτητα διαπιστευτήρια θα πρέ... Επίσης πιστεύουμε ότι οι μακροχρόνιες επενδύσεις θα πρέπει να ε, παρακάμπτουν τους κινδύνους Forex και RAN και επίσης ε, ότι θα πρέπει να γίνονται και διάφορες ε, δοκιμές οι οποίες να αφορούν τους πραγματικούς κινδύνους και όχι τίποτα περίεργους στόχους fancy objectives λέει ο μιλητής. έτσι ώστε να υπάρξει στήριξη της πραγματικής ε, ε, οικονομίας. Ε, θα πρέπει να βάλουμε κάποια ποσοστά της 100 και αυτό είναι καλή ιδέα ότι η επένδυση σε real assets θα πρέπει να γίνεται μονάχα εάν μπορεί να επιτρέψει την ευκολότερη ροή κεφαλαίου. Όπως και ο Ζαμπόλ έλεγε θα πρέπει να είναι μακροχρόνια. Μας απασχολεί, μας προβληματίζει λίγο ε, το, η δυνατότητα άρσης ε, των ε, κανόνων και εκεί γίνεται αναφορά στα πέντε χρόνια. Έχουμε τη, λοιπόν την τροπολογία 2.12 η οποία αναφέρεται στο θέμα αυτό. Επίσης αυτό που δεν καταλαβαίνουμε ε, είναι γιατί η ε, Κομισιόν ε, δεν αναφέρεται σε νόμους οι οποίοι είναι ταυτόσιμοι με τους νόμους του IMF. Καταθέτουμε τροπολογίες και κατά αυτή την έννοια. Τέλος, βλέπουμε ένα πρόβλημα με το listing γιατί κατά την άποψή μας δημιουργεί ένα πρόβλημα διαχείρισης με, άλλους, με, άλλα λόγια εμείς ε, πιστεύουμε ότι οι αγορές και ε, τα, τα, stock markets change δεν είναι μακροχρόνια θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσον μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά εν πάση περιπτώσει είναι κατατεθειμένες οι τροπολογίες μας. Ε, ε, δεν θα συμφωνήσουμε επίση ε, και με αυτά που λένε οι Ντεμπάκερ και Λούλινγκ όσον αφορά την άμεση διόρθωση της θέσης. Υπάρχει η 2015 του Ζαν Πολ ε, σχετικά με την συμμόρφωση των, ε, προς τα κριτήρια ε, και για δύο χρόνια συμφωνώ. Επίσης για το τέλος του κύκλου ζωής, end of life και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος. Έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά κάποιες άλλες τροπολογίες, κυρίως με τις τροπολογίες οι οποίες ε, δεν θέλουν να επιτρέψουν ε, την επένδυση από λιανικούς ε, επενδυτές. Να μην μπερδεύουμε εδώ τους στόχους. Εμείς θέλουμε τον καλύτερο τρόπο επένδυσης των λιανικών επενδυτών και λέμε ότι αυτός είναι μέσω των users funds που λειτουργούν καλά, υπάρχουν, αφορούν ή στοχεύουν στους λιανικούς επενδυτές και βεβαίως ε, τα users funds μπορούν να επενδύσουν σε LTIFs. Δεν έχει έννοια να βάλουμε όλους ε, τους ε, δυνατούς ελέγχους στην ρύθμιση LTIFs. Νομίζω ότι ο δρόμος των users funds είναι καλύτερος δεν καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση ή δικαιολογία για χαλάρωση των ε, κανονισμών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος λόγος ε, και αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 207 συγκεκριμένα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα στην αγορά τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν ε, τους πάντες. Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ε, να μπερδέψουμε, να αλλάξουμε την, ε, τον κανονισμό ΕΛΤΙΦ. E Επίσης, η δυνατότητα διαχείρισης του ΕΛΤΙΦ χωρίς επιπλέον ε, πρόνοια και ε, το θέμα των ε, αρμοδίων αρχών. Ναι, λέμε ότι έχουμε υποβάλει μια τροπολογία σχετικά με τις με τους μελλοντικές εκτιμήσεις μας. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Uh, Ευχαριστώ. Στον κατάλογο έχω τον Ζαν Πολ και την Αστρίτ Λούλινγκ. Νομίζω ότι θα προλάβουμε διότι η Astrid Λούλινγκ πρέπει να φύγει, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στην Άστρι... στον Ζων Πολ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικές παρατηρήσεις μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Ρόδη για την τόσο καλή συνεργασία. Επειδή ε, έκανε ένα ερώτημα θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ο στόχος δημιουργίας αυτών των κεφαλαίων είναι πάρα πολύ χρήσιμος, αξιέπαινος και διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα μακροπρόθεσμη χρηματοδότησης. Έχω κάνει τροπολογίες για διάφορα θέματα, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, στις εισηγμένες εταιρείε, ε, ε, πρόθεση των επενδύσεων στην Ευρώπη, να έχουμε διαχείριση χαρτοφυλακίου αποτελεσματική, συμπλήρωση του κανονισμού για διοικητικές κυρώσεις και επιβολή τους και έρχομαι στο ερώτημα που έκανε προηγουμένως η κυρία Κράτσα, τη δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Γιατί κάνω αυτή την πρόταση. Απλούστατα, διότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου να είναι κλειστά αυτά τα κεφάλαια για ένα συγκεκριμένο διάστημα και μετά να φανεί σκόπιμο ε, να γίνει ενδεχομένως μείωση του κεφαλαίου του ταμείου αυτού με διανομή μετά ε, από την εξαγορά των μεριδίων εκείνων που θέλουν να αποχωρήσουν από το δυτικό κεφάλαιο. Δεν ξέρω, το ξέρω ότι θα υπάρχουν κανόνες και πλαισίωση, αλλά να μην απαγορεύσουμε αυτή την ε, ευελιξία ε, που μπορεί να επιτρέπει κάποιες ε, προσαρμογές όταν έχει μια δεδομένη οικονομική κατάσταση ένας επενδυτής. Αυτά κατά τα άλλα εμπιστεύω με την εισηγήτριά μας και την κοινή συνεδρίαση των σκιωδών για να βρούμε καλές λύσεις σε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Άστριτ Τλούλινγκ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή δεν θα ήταν άχρηστο να υπενθυμίσουμε ότι ο στόχος αυτών των ευρωπαϊκών μακροπροθέσμων επενδυτικών κεφαλαίων είναι να βρεθούν κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν έργα που να ε, είναι προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Όπως γνωρίζουμε, τα κεφάλαια αυτά εξορισμού έχουν μακροπρόθεσμη πρόπτικη πράγμα που τα καθιστά ε, από τη φύση τους κάπως βαριά. Θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία οι επενδυτές να αποζημιώνονται πριν το τέλος ε, του κύκλου ζωής. Αυτό φαίνεται όμως αντιφατικό. Η εμπειρία μας στο παρελθόντος μας έδειξε με διάφορα ε, κεφάλαια ε, ακινήτων Σε περίπτωση μαζικής επιθυμίας αποχώρησης, αυτό αποτελεί κίνδυνο για την ίδια την επιβίωση του επενδυτικού κεφαλαίου και των επενδυτών. Και οι τελευταίοι που θα ζητήσουν να επιστραφούν τα χρήματά τους, τελικά ε, θα είναι χαμένοι της υπόθεσης, τα λεγόμενα κορόιδα. Το ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι με αυτό, αλλά σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προστατεύονται οι επενδυτές. Και με ένα πνεύμα συμβιβασμού με το πρώτο σημείο θα μπορούσαμε ενδεχομένω να σκεφτούμε το εξής. Να περιορίσουμε τους μικροεπενδυτές, τους λιανικούς, σε κάποιους πιο έμπειρους επενδυτές και εύρωστους οικονομικά έτσι ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό το κίνδυνο ρευστότητας. Παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα κατόφλι, ένα ελάχιστο όριο, δεν ξέρω, 5.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Θα το δούμε αυτό στο ε, ε, EUSF και EUSF και μία γραπτή δήλωση και υπογραφή ότι αναλαμβάνω ένα κίνδυνο τον οποίο έχω αντιληφθεί και κατανοώ όταν μπαίνω σε αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο οι συνάδελφοι Χιούμπνερ, Ντεπάκερ, Μόζα, Σιλβί Γκουλάρ, Όλε Σμιτ, Τόμα Μαν, Μπάλτ και άλλοι αναφέρονται επίση σε τέτοια κριτήρια. Επίσης θα επιθυμούσα να υπογραμμίσω ότι τα επενδυτικά κεφάλαια αυτά ονομάζονται ευρωπαϊκά και έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή αγορά επενδυτικών κεφαλαίων και μάλιστα μακροπρόθεσμων και μέσω ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Το να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες τώρα ως προς την κυκλοφορία στην αγορά ε, τέτοιων προϊόντων προς τους ε, λιανικούς επενδυτές αντιτίθεται με το στόχο αυτό και τη φιλοδοξία των κεφαλαίων. Και οι τροπολογίες 278, ε, 123 και 80 κατά την άποψή μου είναι προβληματικές. 80, 123, 278 επίσης και αυτές που έχουν να κάνουν με τη ε, διανομή των κερδών, των μερισμάτων, ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διανομής του κεφαλαίου αυτού και ε, μάλιστα και του αρχικά επενδεδημένου κεφαλαίου. Στόχος των κεφαλαίων αυτών είναι να αυξηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια για να μπορούν να χρηματοδοτούνται μακροπρόθεσμα έργα θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα ένα εναλλακτικό επενδυτικό κεφάλαιο να μπορεί να χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό επενδυτικό κεφάλαιο Μακροπρόθεσμο. Αυτό ενδεχομένως θα επέτρεπε εγκάρσιες επενδύσεις και οικονομίες κλίμακος καθώς επίσης και διαφοροποίηση έτσι ώστε να ανταποκριθούμε με τρόπο αποτελεσματικό στον πρώτο και πρωταρχικό μας στόχο. Τέλος, για να μπορέσουν να συλλεγούν κεφάλαια για τα έργα αυτά, δεν θα πρέπει να απαγορεύεται να επενδύει κανείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε να επιβάλλουμε κοινωνικούς στόχους ή οικολογικούς φερρυπίν αυστηρούς, γιατί έτσι θα περιορίζεται η δυνατότητα επενδύσεων. Διαφωνώ λοιπόν με τους πρασίνους επ' αυτού. Αυτοί οι περιορισμοί θα απεθάρρυναν ε, πολλούς ε, φορείς και παράγοντες της αγοράς από την ίδια τη δημιουργία τέτοιου ε, κεφαλαίου τον ΕΜΕΚ, άλλο ακρονίμιο που θα πρέπει να θυμόμαστε, Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια. Και στο ίδιο πνεύμα, κανονικά θα πρέπει ε, να μας ενδιαφέρει να επιτύχει η νομοθεσία αυτή στην πράξη. Και γι' αυτό και εγώ και άλλοι συνάδελφοι προτείναμε να υπάρχει η δυνατότητα για ένα τέτοιο επενδυτικό κεφάλαιο να μπορεί να επενδύει ε, αμέσως ή σε συγκεκριμένες αξίες με εναλλακτικούς τρόπους επενδύσεων με ειδικά στοιχεία ενεργητικού και ειδικέ δομές αλλά όπου να είναι κάθε φορά ε, ένα συγκεκριμένο επιλέξιμο ενεργητικό. Έχω αυτές τις ανησυχίες και σας τις ε, αναφέρω. Για να μπορέσουν να πετύχουν τα επενδυτικά αυτά κεφάλαια χρειάζεται ε, προσοχή. Και να λάβουμε υπόψη αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χρόνο και είναι παρούσα η Κομισιόν. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην Κομισιόν. Παρακαλώ, Τίλμαν. Ναι, πολύ σύντομα. Τα συνηθισμένα τρία σημεία τώρα όμως συνδέονται μεταξύ τους. Ακούσαμε πολλά για τις ε, δυνατότητες ανάκτησης ε, για όλους, για κάπου ή για κανένα. ή για κανέναν, ε, επέκταση της διάρκειας ζωής, και, τις, και την ε, εισαγωγή. Και το θέμα είναι ότι, και το σκεφτήκαμε πολύ αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολοκλήρου και το σκύλο χορτάτο. Δεν μπορεί κανεί ε, να είναι μακροπρόθεσμο επενδυτή ε, και να έχει δυνατότητε ανάκτηση βραχυπρόθεσμε. Αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ του και συμφωνώ ότι τα, ε, ε, τα κεφάλαια ε, ακινήτων με απεριόριστη προθεσμία στο τέλος το έχουν αποδείξει αυτό. Εξετάζουμε λοιπόν τις προτάσεις σχετικά με τον κύκλο ζωής μπορεί να τροποποιηθεί. Έτσι λοιπόν μπορεί το ε, ταμείο να συνεχίσει να υπάρχει, το κεφάλαιο να συνεχίσει να υπάρχει, δεν χρειάζεται να εκαθαριστεί, αλλά θα πρέπει να συμφωνηθεί η ανάκτηση από όλου του επενδυτέ. Ε, και όσοι θέλουν να το κάνουν αυτό ε, με τη λήξη της προθεσμίας θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν αυτό. Ε, κατά τα άλλα όμως ε, έχουμε τον ε, κύκλο ζωής. Μπορεί να υπάρξει νέος κύκλο ζωής εφόσον υπάρξει συμφωνία. Πιστεύουμε όμως ότι η εισαγωγή σε δευτερεύουσα αγορά του κεφαλαίου είναι χρήσιμο εργαλείο για να αυξηθεί η ρευστότητα για τους επενδυτές χωρίς να επιβαρυνθεί ο διαχειριστής με πρόορια ανάκτηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Μπορεί λοιπόν ο επενδυτής να μπορεί να βρει αγοραστή στην δευτερογενή αγορά και είμαστε υπέρ αυτού και θα εξετάσουμε τις ανησυχίες του Φιλίπ Λαμπέρ, το ότι υπάρχουν γενικά βραχυπρόθεσμοι οριγορές, θα το κοιτάξουμε αυτό. Είμαστε όμως υπέρ της ε, εμπορίας της δευτερογενής αγοράς, διότι αυτό σημαίνει ότι έτσι δεν κυμαίνεται συνεχώς η βάση των επενδυτών για τον διαχειριστή. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ε, είχα εφεύρει το retail repo. Ε, είναι μια ιδέα την οποία είχα παρουσιάσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, πάντως είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Να προσπαθήσουμε έτσι να προσελκύσουμε περισσότερους στις ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις πρόκειται για μια, περίπτωση, για μια ε, ε, επιλογή σε περίπτωση επιδούσα ανάγκη. Ε, υπάρχει κανεί άλλο που θέλει να πάρει το λόγο. Εάν όχι, να δώσω το λόγο πάλι στην εισηγήτρια. Ρόδη, παρακαλώ. Κυρία Κράτσα. Κυρία Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, διότι αφενό φαίνεται πώ όλοι ε, συνειδητοποιούμε τη σημασία που έχει το εγχείρημα, αφετέρου δεν έχουμε μεταξύ μας αποκλίνουσες προσεγγίσεις, προβληματισμοί και τεχνικές προσαρμογές πρέπει να γίνουν. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε ε, σε μια συμβιβαστική πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, για την πρόταση που έχει υποβάλει και τη συμπαράσταση που μας έχει κάνει στην επεξεργασία όλων αυτών των θέσεων και την ε, ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η συγγήτρια, θα ψηφίσουμε, έχουμε στόχο στις 17 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή, για να πάμε μετά στην Ολομέλεια του Απριλίου. Άλλη πολύ βαριά ολομέλεια αυτή. Αυτά. Στα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 3 το απόγευμα. Μέχρι τις 6.30. Ευχαριστώ πολύ και χαίρετε.